Good, meine... Ο πρόεδρος Λάνγκε. κάρλος. Λοιπόν, κυρίε και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση και επισήμω, πρόκειται για την ακρόαση ιδίω για τις γενικευμένες προτιμήσεις ΣΥΝ που ε, έχει, δηλαδή η σχετική νομοθεσία έχει ήδη μια ηλικία δύο ετών και επιθυμούμε να εξετάσουμε που χρήζει βελτιώσεως. Ε, Είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένο γιατί κοντά μας βρίσκονται γνώστες του θέματος, εμπειρογνώμονες. Πρώτα βεβαίως η Σεσίλια Μάνστρομ, η Επίτροπος Εμπορίου. Βεβαίως και ο Κρίστιαν Λέφλερ που είναι αναπληρωτής διευθυντής της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικών Δράσεων. Καλώς ήρθατε και εσείς κύριε Λέφλερ από το GSP Plus προτιμήσεις δηλαδή έχουμε δύο χώρες οι οποίες επωφελούνται από αυτά τον κύριο Ασούφ Αλή που είναι Special Assistant του Πρωθυπουργού του Πακιστάν βρίσκεται λοιπόν κοντά μας και το πρόσωπο αυτό και ο κύριος Ντόρι που είναι πρέσβης της Μογγολίας παρά τη Ευρωπαϊκή Ενώση. Σας καλωσορίζω και εσάς. Το δεύτερο μέρος θα ασχοληθεί περισσότερο με την εφαρμογή και ένταξη στον μηχανισμό GSP Plus της κοινωνίας των πολιτών. Εκεί θα έχουμε τη χαρά να καλωσορίσουμε τέσσερις εμπειρογνώμονες. Την κυρία Βάργα, Διευθύντρια του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας, Βέγγλερ από το ε, Smith Association, τον κύριο Ρέινι, συντονιστή του οργανισμού Justice and Peace και τον κύριο Άβαν, πρόεδρο της Πακιστανικής Ομοσπονδίας Εργαζόμενων. Ευχαριστώ λοιπόν όλα τα πρόσωπα αυτά για την παρουσία τους εδώ και φαίνεται πράγματι ότι θα είναι ή μάλλον είναι μια ομάδα ε, ανθρώπων με εντυπωσιακή εμπειρία και γνώση. Χαίρομαι επίσης που βλέπω και έναν αριθμό συναδέλφων της Διευθύνουσας Επιτροπής της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου που επιθυμούν να παρακολουθήσουν την συζήτηση αυτή για τις γενικευμένες προτιμήσεις γιατί βέβαια είναι κρίσιμο θέμα και για πολλά μέλη του ΠΟΕ. 20 περίπου μέλη της Διευθύνουσας Επιτροπής από Ρωσία, Ιορτανία, Ινδονησία, Κολομβία, Μποτσουάνα, Κίνα και Ινδίες και βεβαίω και από Ευρωπαίους, ε, συγνώμη, από Ευρωπαίους εταίρους. Καλώς ορίσατε λοιπόν και εσείς όλοι. Η νομοθεσία GSP, Κοινοβουλίου και Συμβουλίου δηλαδή, όπως είπα, έχει ήδη αρχίσει να εφαρμόζεται εδώ και μια διετία. Στόχος μας είναι να αναλογιστούμε αν αυτό είναι και το σωστό εργαλείο για την εφαρμογή των 27 συνθήκων ή συμβάσεων που συνδέονται με την ομοθεσία αυτή. Γιατί έχουμε και περιορισμένο χρονικό ορίζοντα της τάξης των 10 ετών. Και θέλουμε να δούμε λοιπόν πώς θα πρέπει να προχωρήσουμε. Αυτός είναι και ο λόγος που χαίρομαι που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει κάνει σχετική έκθεση. Η δε Επίτροπος κυρία Μάλμστρομ θα αναπτύξει τα εκθέσεις αυτής. Επιθυμώ να δώσω το λόγο και στην κυρία Σερά, ωστόσο, που είναι της Νομικής Επιτροπής για να σας απευθύνει χαιρετισμό. Καταρχήν, θα ήθελα να πω ότι χαίρομαι που μπορούμε να θίξουμε αυτό το εγκάρσιο θέμα που άπτεται αρμοδιοτήτων Ιντα Κέντροα και ελπίζω να είμαστε αποτελεσματικοί θα πρέπει να τονίσουμε τη σημασία της εμπορικής πολιτικής και των μέσων που έχουμε στη διάθεσή μας για να επηρεάσουμε τα παγκόσμια δεδομένα, ιδιαίτερα την εφαρμογή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων παγκοσμίω. Έχουμε ελοένα και περισσότερες κρίσεις και μέσα στα πλαίσια των γενικευμένων προτιμήσεων το σύστημα αυτό θα πρέπει να διέπει τη σκέψη μας ως προς την εξωτερική μας δράση και τις σχέσεις με τρίτες χώρες. Μέσω του διεθνούς εμπορίου μπορούμε να δημιουργήσουμε ευεργετικές εμπορικές σχέσεις, αλλά θα κάναμε μεγάλο ε, λάθος εάν δεν συνοδεύσουμε αυτές τις πολιτικές ε, με μέτρα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ε, εργασιακών δικαιωμάτων, προστασία του περιβάλλοντος και αντιμετώπισης των κλιματικών αλλαγών μέσα στα πλαίσια της Ατζέντα 2030. Θα θέλαμε λοιπόν να ακούσουμε τους εμπλεκόμενους φορείς για να δούμε ποια είναι η οικονομική χρησιμότητα αυτού του συστήματος και οι σχέσεις μεταξύ εμπορίου και ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Πρόκειται για κοινό μας συμφέρον να υπερασπιστούμε τη δημοκρατία και την πρόοδο. Βεβαίως κάθε ευεργετούμενη χώρα μπορεί να έχει διαφορετική, λίγο διαφορετική θεώρηση, αλλά 27 διεθνείς συμβάσεις θα πρέπει να έχουν καθολική εμβέλεια. και αυτό έμπρακτα ο πρόεδρος Λάγκε έθεσε πολύ σημαντικά ερωτήματα δύο χρόνια μετά τη θέση εφαρμογή του νέου κανονισμού θα πρέπει να δούμε κατά πόσο είναι το καταλληλότερο μέσο και πώς μπορούμε να συνεχίσουμε με τις δεσμεύσεις μας. Επίσης, πώς μπορούν να είναι αποτελεσματικά τα μέτρα του κανονισμού, άρθρο 15, όταν τα πράγματα δεν πάνε όπως θα θέλαμε και να αναστείλουμε τις γενικευμένες προτιμήσεις. Επίσης, πώς οι τοπικές αρχές και εθνικές αρχές θα μπορούσαν να παρεύουν πιο διαρθρωμένα. Η Επιτροπή θέλει να ε, συνεχίσει τις επαφές με την κοινωνία των πολιτών. Σήμερα κάνουμε έναν απολυσμό της διετίας αυτής και ελπίζω να βρούμε στοιχεία έτσι ώστε όλοι να μπορέσουμε να βελτιώσουμε αυτό το πλαίσιο. Από την Υποεπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων θα συνεργαστούμε με την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου προς αυτή την κατεύθυνση. Ο Πρόεδρος Λάγκη, σας ευχαριστώ πολύ. Μια πρακτική υπόμνηση έχουμε περιορισμένο χρόνο. Βεβαίως θέλουμε να ακούσουμε όλους τους ειδήμονες και όλες τις ειδήμονες και να μπορέσουμε να διεξαγάγουμε και συζήτηση. Γι' αυτό θα σας παρακαλέσω όλες και όλους να προσέξετε ιδιαίτερα τα όρια του χρόνου αγόρευσης. Έχουμε δώσει 7 λεπτά στον καθένα και στην καθεμία σε Σίλια Μάλμστρομ. Ορίστε λοιπόν έχετε το λόγο κυρία μου. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και εσάς κυρία Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι ευχαριστώ το Κοινοβούλιο που οργανώνει την παρούσα ακρόαση. Έχει μεγάλη σημασία το θέμα αυτό. Γνωρίζετε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εγώ προσωπικά αποδίδουμε μεγάλη σημασία στη διασύνδεση μεταξύ εμπορίου και ευρωπαϊκών αξιών όπως τα ανθρώπινα δικαιώματα, η βιώσιμη ανάπτυξη και τα βάζουμε στο επίκεντρο των προσπαθειών μας. Μάλιστα αυτά τα εξηγήσαμε και στην ανακοίνωσή μας του περσινού χρόνου. Επειδή η σημασία ε, της υπόθεσης αυτής γίνει ακόμα μεγαλύτερη με το χρόνο που περνά και μάλιστα και εν του μεταναστευτικού, εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει εργαλεία που μπορούν να συμβάλλουν στην ανάπτυξη των αναπτυσσόμενων χωρών, πρέπει να τα χρησιμοποιήσουμε και μας τα χρησιμοποιήσουμε καλύτερα. Το πρόγραμμα SIN, το Γενικευμένο Σύστημα Προτιμήσεων δηλαδή, έχει σήμερα μεγαλύτερη σημασία από ποτέ. Προβλέπεται προβλεπόταν για το 2014-2015 για 15 αρχικά χώρες. Συνολικά στον πληθυσμό των πολλών εκατομμυρίων 30% ε, ήταν νέοι. Χρειάζεται λοιπόν να κατανοηθεί ο τρόπος με τον οποίο το εμπόριο μπορεί να συμβάλλει στην ανάπτυξη του βιώσιμου εμπορίου και της βιώσιμης ανάπτυξης, δίνοντας στους εταίρους μας από τις χώρες αυτές πρόσβαση σε μια πολύ μεγάλη αγορά, βελτιώνοντας έτσι και την ε, ευημερία τους. Πρόσβαση και υπόσχεση προς τις κυβερνήσεις, μάλλον υπόσχεση από τις κυβερνήσεις τους να εφαρμόσουν 27 συνολικά διεθνείς συνθήκες για ανθρώπινα δικαιώματα, εργατικά δικαιώματα, ε, βιώσιμη ανάπτυξη καθώς και ε, χρηστή διακυβέρνηση. Έτσι λοιπόν έχει το δυναμικό να δημιουργήσει έναν ενάρετο κύκλο να προωθήσει την οικονομική ανάπτυξη. Η οικονομική ανάπτυξη διευκολύνει βεβαίω και την εφαρμογή των διεθνών συνθήκων. Γίνονται ανοιχτέ οι κοινωνίε που αυτό επίση οδηγεί σε μεγαλύτερη ευημερία και περισσότερε επενδύσει. Αυτά που συζητούμε σήμερα εδώ λοιπόν είναι η πρώτη έκθεση σχετικά με το πώ αποδίδει η προσπάθεια αυτή στην πράξη. Τον προηγούμενο μήνα μαζί με την κυρία Μογκερίνη εκδώσαμε την πρώτη έκθεση του προγράμματος GSP Plus και του γενικότερου προγράμματος γενικευμένων προτιμήσεων. Δύο χρόνια μετά από τη θέση του σε εφαρμογή. Η έκθεση έχει μεγάλη σημασία ως εργαλείο. Για πρώτη φορά η Ευρωπαϊκή Ένωση συστηματικά και επισήμως λαμβάνει θέση επί των προσπαθειών των εταίρων μας για τη βελτίωση όλων αυτών των παραμέτρων που ανέφερα προηγουμένως. Θα πω λοιπόν λίγα λόγια για αυτό. Αυτά που λέει η έκθεση και αυτά που δεν λέει. Η έκθεση δίνει μια ξεκάθαρη εικόνα της σημερινής πραγματικότητας στην προσπάθεια εφαρμογής των 27 core conventions, βασικών αυτών συνθήκων. Αλλά και σημειώνει και τι χρειάζεται ακόμη για να επιτευχθεί πρόοδος και τώρα και στο μέλλον. Για παράδειγμα, Πακιστάν και παιδική εργασία. Ο κύριος Άλλη, ελπίζω να συμφωνήσει όταν θα μιλήσει αργότερα, ότι η εργασία των παιδιών είναι σημαντικό και βαρύ, τραγικό πρόβλημα σε πολλές περιοχές της χώρας του. Όμως, οι επαρχίες στο Πακιστάν καταβάλουν προσπάθεια για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα αυτό. Έχουν ήδη ε, ψηφιστεί νόμοι, έχουν ήδη διατεθεί κονδύλια για να αυξηθούν οι επιθεωρήσεις εργασίας στο Πουντζάμπι, άλλο τμήμα του Πακιστάν μάλιστα έχει προωθηθεί στην τοπική κοινοβουλευτική συνέλευση. Αναμένουμε βεβαίως να, να ληφθούν και άλλες δράσεις και στην επαρχία ΣΥΜΤ και στο Βελουχιστάν. Άλλο πρόβλημα τώρα, άλλο ε, παράδειγμα μάλλον της Μογγολίας. Είμαι βεβαία ότι θα χαρεί ο πρέσβης της Μογγολίας που θα δει στην έκθεση ότι αναφέρεται ότι η κυβέρνησή του έχει αναλάβει τη δέσμευση να προωθήσει τα ε, θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα στην Μογγολία. Σημειώνω επίση έστω και αν δεν περιλαμβάνεται άμεσα στο GSP Plus ότι η Μογγολία κατάργησε την θανατική ποινή. Και εδώ υπάρχει χώρος για βελτιώσει, ωστόσο. Δηλαδή θα πρέπει η Μογγολία να καθιδρύσει έναν μηχανισμό για την εξέταση καταγγελιών για βασανιστήρια και κακομεταχείριση. Άλλο παράδειγμα, Αρμενία. Εκεί η κυβέρνηση έχει εγκρίνει σχέδιο στρατηγική κατά τη διαφθοράς που να, που να ε, περιλαμβάνει όλους τους τομείς από την αστυνομία μέχρι την έσπραξη φόρων. Βεβαίως η διαφθορά εξακολουθεί να παραμένει μεγάλο πρόβλημα. Αυτή η νομοθεσία αντιδιαφθοράς πρέπει βεβαίως να βελτιωθεί και να εφαρμοστεί με τον δέοντα τρόπο. Τονίζω επίσης ότι η Αρμενία καλείται να καταβάλει ε, προσπάθειες και να επιτύχει πρόοδο και στο εκλογικό της σύστημα. Για κάθε μία από τις χώρες εταίρους λοιπόν γίνεται μια σε βάθος ανάλυση των επιτευγμάτων τους. Αυτά που δεν θα βρείτε ωστόσο στην έκθεση είναι τα εξή. Είναι μια κατάταξη των χώρων, διότι κάτι τέτοιο δεν ανταποκρίνεται στην περιπλοκότητα των ζητημάτων. Όλες οι χώρες καταβάλουν προσπάθειες για να εκπληρώσουν τους στόχους του συστήματος GSP-SYN και γι' αυτό δεν κάνουμε συστάσεις να αποσυρθούν να αφαιρεθούν δηλαδή οι γενικευμένες προτιμήσεις για κάποια χώρα, διότι γνωρίζουμε ότι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε είναι περίπλοκα, είναι από μακρού χρόνου υπαρκτά και εμείς δεν έχουμε λύσει όλα τα προβλήματά μας μέχρι και εδώ, μέχρι και η δεκαετία του 80 η παιδική εργασία και σε χώρες μέλη της Ένωσης ήταν μια πραγματικότητα. Χρειάζεται λοιπόν να δώσουμε μακροπρόθεσμη ενίσχυση στις χώρες εταίρους και γι' αυτό προβλέπουμε δεκαετή ορίζοντα για μακρού χρόνου λοιπόν εμπλοκή. Το ίδιο είναι μακροχρόνιες και οι δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει οι κυβερνήσεις των χωρών εταίρων. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι όποιος θέλει κάνει ό,τι θέλει. Εξετάζουμε συγκεκριμένα στην έκθεση που πρέπει να σημειωθεί πρόοδος και στον διάλογο που διεξάγουμε με τις κυβερνήσεις των χωρών αυτών. Στη βάση ερωτηματολογίου που αποτελεί και ένα βαθμολόγιο στο τι πρέπει να πράξει κάθε μια κυβέρνηση δηλαδή για να βελτιώσει την κατάσταση επιτόπου. Οι δε εταίροι μας αντιλαμβάνονται τη σημασία του διαλόγου και αυτή την παρακολούθηση monitoring. εμεί, η Ευρωπαϊκή Ένωση, θα συνεχίσουμε να ασκούμε πίεση μέσω του διαλόγου αυτού και θέλουμε να δούμε πραγματικέ προόδου. Το σύστημα GSP Plus δεν σημαίνει ότι πρέπει να παραμείνουν εκεί που ήταν όταν, όταν εντάχθηκαν στο σύστημα αυτό οι χώρες πρέπει να συνεχίσουν να προχωρούν. Στην επόμενη έκθεση monitoring θα εξετάσουμε προσεκτικά να δούμε πού επιτεύχθηκαν βήματα πρόοδου σε όλες τις χώρες και σε αυτές που εκπροσωπούνται σήμερα εδώ. Και βεβαίως οποιαδήποτε υποχώρηση, οπισθοδρόμηση δεν είναι επιλογή γιατί μπορεί να αφαιρεθούν οι προτιμήσεις από τις συγκεκριμένες χώρες όπως κάναμε για την Μιανμάρ, για τη Σιριλάνκα και για τη Λευκορωσία στο παρελθόν και είμαστε διατεθειμένες να το πράξουμε και στο μέλλον. Επανέρχομαι ωστόσο στην αφετηρία. Ο βασικός στόχος του προγράμματος είναι να φτιάξει, να στήσει τα πόδια του έναν ενάρετο κύκλο και γι' αυτό συνεργάζεται τόσο στενά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την Υπηρεσία Εξωτερικών Δράσεων και θα ακούσουμε πολύ σύντομα τώρα τον ε, ε, διευθυντή της Θέλουμε όμως να εργαστούμε ακόμα πιο στενά μαζί με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, που ο ρόλος του είναι σημαντικός, διότι εσείς οι Ευρωβουλευτές έχετε τις επαφές σας, έχετε επαφές με τους ε, κοινοβουλευτικούς συναδέλφους σας στις χώρες αυτές, ταξιδεύετε, βλέπετε τα πράγματα επί τόπου, μπορείτε να ενθαρρύνετε τις χώρες αυτές να σημειώσουν πρόοδο, ερχόμενοι σε επαφή με την κοινωνία των πολιτών και ασκώντας πίεση και εσείς για να ε, σημειωθούν βήματα πρόοδου. Ελπίζω λοιπόν ότι θα μπορέσουμε να συνεργαστούμε χέρι με χέρι για την επίτευξη ακόμη καλύτερων αποτελεσμάτων. Και ελπίζουμε συν το χρόνο να βελτιωθεί και η συνεργασία, εκφράζουμε αυτή την ελπίδα εμείς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μια πιο στενή συνεργασία δηλαδή με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και εσάς κυρία Πρόεδρε. Ο Πρόεδρος Λάγκη, σας ευχαριστώ πολύ για την εισαγωγή. Θα δώσω τον λόγο στον κύριο Άλλη του Πακιστάν. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, μέλη της Επιτροπής, εκπρόσωποι της Κοινωνίας των Πολιτών, κυρίες και κύριοι, είναι μεγάλη τιμή να απευθυνθώ σε αυτή την έγκριτη Επιτροπή του Ευρωκοινοβουλίου για το θέμα αυτό του συστήματος GSP-SYN η δημόσια αυτή ακρόαση είναι μια χρήσιμη ευκαιρία για να καταγράψουμε την πρόοδο που έχει επιτελεστεί από το Δεκέμβριο του 2014 και μαζί με το Ευρωκοινοβούλιο να εντοπίσουμε τα προβλήματα και τις ελλείψεις καθώς και πώς πρέπει να προχωρήσουμε. Θα αξιοποιήσω αυτή την ευκαιρία για να μιλήσω για τις σχέσεις του Πακιστάν με την Ευρωπαϊκή Ένωση, σχέσεις που έχουν ενδυναμωθεί σε πολλούς τομείς ανυπομονούμε από το εμπορικό επίπεδο να περάσουμε σε πιο στρατηγικά θέματα στη συνεργασία μας αυτή. Κύριε Πρόεδρε, το Πακιστάν έχει προχωρήσει πολύ από τις εκλογές του 2013. Η πραγματικότητα στο Πακιστάν εντωμεταξύ έχει αλλάξει. Το Πακιστάν είναι μια χώρα όρημη και δημοκρατική, που λειτουργεί εύρυθμα. Η ασφάλεια έχει βελτιωθεί η σταθερότητα υπάρχει. Υπάρχει σημαντική αντιμετώπιση της τρομοκρατίας σε δύσκολες στιγμές για τον κόσμο. Ε, η Ευρώπη ανησυχεί βεβαίως ακόμη για το τι συμβαίνει. Ε, άρχισαν σχετικέ επιχειρήσεις το 2014 και υπάρχει πρόγραμμα δράσης από τον Ιούνιο του 2015 με σοβαρές ε, επιτυχίες. Υπάρχει λοιπόν αίσθηση ανακούφιση και ηρεμία σε όλη τη χώρα. Με περισσότερη οικονομική σταθερότητα. Φαίνεται σαν να έχουν περάσει δύσκολη κυρία για το Πακιστάν και να βελτιώνονται οι οικονομικέ συνθήκε. Δυστυχώ όμω αυτή η μεταβαλλόμενη πραγματικότητα του Πακιστάν δεν ε, απηχείται από τα μέσα μαζική ενημέρωση και υπάρχουν και κάποιε θλιβερέ εξαιρέσει. Είναι και το μεγαλύτερο θύμα τη τρομοκρατία του Πακιστάν. Η τρομοκρατία και ο εξτρεμισμό ε, σοβούν. Η οδή ε, το τρομοκρατία. της τρομοκρατίας ε, περνούν από το Πακιστάν. Έχουμε χάσει πάνω από 150 δις ε, δολάρια λόγω των πολεμικών συγκρούσεων και ε, πολλούς πολίτες, πολλές ζωές έχουν χαθεί. Για δεκαετίες είχαμε τέτοια προβλήματα και επειδή η ανθρωπιστική βοήθεια φθήνει από τη διεθνή κοινότητα ε, αντιμετωπίσαμε και πολλές φυσικές καταστροφές μόνοι μας, με πολλές κοινωνικές συνέπειες η καθεμία. Κύριε Πρόεδρε, παρά τις προκλήσεις και τα προβλήματα αυτά, παραμένουμε σταθεροί. Δεν υπάρχει περιθώριο για εσωτερική αμφισβήτηση στο Πακιστάν. Πρέπει να συνεργαστούμε με τους διεθνεί μα εταίρους για να υπάρξει μια συμμετοχική κοινωνία Είναι μεγάλη μας προτεραιότητα για να ε, εφαρμόσουμε αμοιβαίως τους στόχους της ανάπτυξης, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας για το καλό όλων των ανθρώπων του Πακιστάν. Έχουμε ιδιαίτερη μέρημνα για τα δικαιώματα των πολιτών, των μειονοτήτων και των παιδιών και θέλουμε η ευημερία τους να τονωθεί περαιτέρω είναι μέρος συμβαλόμενο όλων των βασικών συνθήκων για τα ανθρώπινα δικαιώματα και των 7 του Πακιστάν σε διεθνές επίπεδο και πρέπει να εφαρμοστούν και στην πράξη και σε επίπεδο κράτους κεντρικού και σε επίπεδο ε, επαρχιών. Υπάρχει ο υπεύθυνο ε, για τον έλεγχο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η υπηρεσία αυτή στο Πακιστάν λειτουργεί ε, χωρίς προβλήματα με μια ευρύτατη εντολή για να παράσχουν την απαραίτητη στήριξη στην κυβέρνηση σε αυτές τις δύσκολες ευθύνες που έχουν να φέρουν πέρας για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Κύριε Πρόεδρε, με μεγάλη ικανοποίηση μπορώ να απευθυνθώ στον, στο σώμα σας και να σας πω ότι το Φεβρουάριο του 2016 ε, εγκρίθηκε το Εθνικό Πρόγραμμα Δράσης για τη βελτίωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την κατάστασή του στο Πακιστάν. Μιλάμε για μια συνολική επισκόπηση ε, όλων ε, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της κατάστασής τους στο Πακιστάν με έξι θεματικές ενότητες και 16 ε, αποτελέσματα στόχους για να πετύχουμε συγκεκριμένα βήματα πρόοδου για τα ανθρώπινα δικαιώματα στο Πακιστάν. Αυτές οι έξι περιοχές είναι πρώτον, ε, το νομικό πλαίσιο ε, και τα ένδικα μέσα. Ξέρουμε ότι αυτά για τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι απαραίτητα προκειμένου να εκπληρώσουμε τις διεθνεί μα υποχρεώσει. Υπάρχουν ε, προβλέψεις για μεταρρυθμίσεις των ε, ισχυών των νόμων και την έγκριση νέων. Επίσης, ε, δωρεάν νομική αρρωγή για τα θύματα παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Δεύτερον, το σχέδιο καθορίζει τέσσερι τομεί προτεραιότητα για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Για μεγάλα μέρη τη κοινωνία, όπω την προστασία των γυναικείων δικαιωμάτων, την προστασία των παιδικών δικαιωμάτων, την προστασία των δικαιωμάτων των μειονοτήτων και όσων έχουν ειδικέ ανάγκες. Τρία. Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί στο σχέδιο για την παιδεία στα πλαίσια των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ώστε να υπάρχει συμμετοχή όλων και μια προοδευτική ολοκλήρωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τέσσερα. Προτινόμενε δράσει για την οικοδόμηση δυνατοτήτων ε, σε περιοχέ συγκεκριμένε με τη συμμετοχή αυτών των επαρχιών και των αρχών του και με καταγραφή των όσων έχουν επιτευχθεί στον κάθε τομέα. Πέμπτο, το Εθνικό Πρόγραμμα Δράσης προτείνει τη δημιουργία και την ενδυνάμωση και την πραγματική λειτουργία των θεσμών που ασχολούνται με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και τελευταίο, αλλά όχι λιγότερο σημαντικό, το πρόγραμμα Προτείνει τη δημιουργία ομάδας κρούσης για την ε, επί, εποπτεία για τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων με συγκεκριμένους μηχανισμούς και τον έλεγχο α, ε, της σωστής δαπάνης των κονδυλίων για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Κύριε Πρόεδρε, για να υπάρξει σωστή εκτέλεση του εθνικού αυτού προγράμματος δράσης πρέπει να προβεθούν και τα ανάλογα κονδύλια για το φετινό δημοσιονομικό έτος που τελειώνει τον Ιούλιο του 2016 και για το επόμενο δημοσιονομικό έτος που ξεκινάει τον Ιούλιο του 2016 και ολοκληρώνεται τον Ιούνιο του 2017. Ευχαρίστω να σα δώσω τι λεπτομέρειε του τεχνικού Προγράμματος δράση για τη βελτίωση τη κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την συγκεκριμένη εκταμείευση κοντιλίων σε όποιον ενδιαφέρεται να τα δει. Έχουμε μια πολύ στενή δέσμευση ε, με όλε τι ειδικέ διαδικασίε και τα υποχρεωτικά εργαλεία που προβλέπονται από τον ΟΗΕ. Πρόσφατα ε, επεκτείναμε ε, την αναφορά που παραδίδεται στον ύπατο εκπρόσωπο του ΟΗΕ για να καλύψουμε και άλλους τομείς, να υπάρξει ευθυγράμμιση και να παρουσιάσουμε το εθνικό μας ε, όραμα και να το εκφράσουμε σε συγκεκριμένα προγράμματα έως το 2025 με τη συμμετοχή των ανάλογων υπηρεσιών και την παροχή συγκεκριμένων δικτύων κοινωνικής προστασίας, την εξάλληψη της φτώχειας και την παροχή όλων των μορφών κοινωνική προστασία. Για μα, Πρόεδρε, το πρόγραμμα GSPC είναι ένα εμβληματικό, ένα ένα εμβληματικό, μια εμβληματική έκφραση, ένα σύμβολο τη στήριξη τη Ευρωπαϊκή Ένωση για το Πακιστάν. Και θέλουμε να δράξουμε όλε τι ευκαιρίε που προκαλεί το σύστημα αυτό για να υπάρξει περισσότερη απασχόληση και για τι νέε γενιέ. Για να αντιμετωπίσουμε τι προκλήσει στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δεν μπορεί να υπάρχουν διακριτικές κυβερνητικές ε, πολιτικές. Θα πρέπει πραγματικά το εμπόριο να βασίζεται σε δημοκρατικά θεμέλια, ελευθερία, δικαιοσύνη και κάτω δικαίου. Γνωρίζουμε τις δυσκολίες, γνωρίζουμε ότι υπάρχει μια διαφορά εδώ, ότι πρέπει να ακολουθήσουμε τη σωστή κατεύθυνση και υπολογίζουμε στη δική σας την στήριξη. Τώρα δίνω το λόγο στον πρέσβη της Μογγολίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Αγαπητοί Πρόεδροι, αγαπητά μέλη της Επιτροπής Διευθύνου Εμπορίου, κυρίες και κύριοι, είναι μεγάλη μου χαρά να είμαι παρόν στην σημερινή ακρόαση και να μιλήσω για την κατάσταση της Μογγολίας ως προς την εφαρμογή του συστήματος ε, γενικευμένων προτιμήσεων. Είναι μέλος η Μογγολία από το 2005. Σήμερα είναι ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος μετά από την Κίνα και τη Ρωσία και συνεισφέραμε για να δημιουργηθούν ευεργετήματα και στους δύο πόλους της συνεργασίας. Όπως ξέρετε υπάρχει άρση των δασμών στην, ε, προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και γι' αυτό μπορούμε να ευεργετηθούμε από το σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων ΣΥΝ. Η έκθεση για την περίοδο 14-15 για τη Μογγολία ως προς τις γενικευμένες προτιμήσεις προβαίνει σε μία έκθεση για τη συμμόρφωση προς τις προδιαγραφές του Σύστηματος Γενικευμένων Προτιμήσεων Plus. Θα καταβάλουμε και περαιτέρω προσπάθειες να ανταποκριθούμε στα κριτήρια και να εποπτεύουμε το πλαίσιο όπως ορίζουν οι 27 συμβάσεις τις οποίες έχουμε προσυπογράψει. Η έκθεση σας δίνει μία συνολική εικόνα της κατάστασης ως προς την εφαρμογή όλων αυτών των συμβάσεων. Δεν θα ήθελα να επαναλάβω αυτές τις δεσμεύσεις, απλώς να σας πω ότι έχουμε καταφέρει εμείς. Ως προς τη Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ε, όπως ξέρετε η Μογγολία έχει υπογράψει όλες τις συμβάσεις και έχει αναλάβει νομοθετικό έργο για να τις εφαρμόσει εθνικά, σε εθνικό επίπεδο. Προσπαθούμε να ενισχύσουμε το σύστημά μας προστασίας ανθρωπίνων δικαιωμάτων με μία ε, ευρεία νομική μεταρρύθμιση με βάση τις 11 συμβάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ως προς την αναθεώρηση του 2015, η αναθεώρηση ήταν επιτυχής. Μετά από την πρώτη έκθεση εμείς Προσυπογράψαμε και το δεύτερο πρωτόκολλο σε σχέση με τα πολιτικά και αστικά δικαιώματα το 2012 καθώς και την προστασία όλων των ε, φυσικών προσώπων, καθώς και το πρωτόκολλο κατά των βασανιστήριων και άλλες ε, μορφές ε, τιμωρίας και την καταδίκη της θανατικής ποινής, καθώς και τα δικαιώματα του παιδιού μέσα στα πλαίσια της ε, διαδικασίας του, του ημερολογιακού έτους του 2014. Τώρα συμμετέχουμε σε εννέα κοινά μέσα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και έχουμε εγκρίνει και τον νόμο για την ισότητα των δύο φύλων, για την ε, καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και αυτό στην περίοδο 2011-2013. Επίσης, θα κινηθούμε ως προς τα δικαιώματα των παιδιών και των ανθρώπων με αναπηρίες. Θα προωθήσουμε και θα υπερασπιστούμε τα ανθρώπινα δικαιώματα. Κατά τη δεύτερη αναθεώρηση, 68 χώρες προέβησαν σε 164 συστάσεις και η Μογγολία δέχτηκε τις 150. Έχει απορρίψει τις 14. Συνεπώς θα ορίσουμε ένα πρόγραμμα δράσης για την εφαρμογή των συστάσεων μετά από διαβούλευση με τις ΜΚΟ, ιδιαίτερα εκείνες που ασχολούνται με το τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Το 2014 προσχωρήσαμε στο δεύτερο πρωτόκολλο σε σχέση με τα αστικά, κοινωνικά και πολιτικά δικαιώματα που στοχεύει στην ε, καταστολή, στην κατάργηση της θανατικής ποινής. Έτσι, η κατάργηση της θανατικής ε, ποινής αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της αναθεώρησης ολοκλήρου του ποινικού δικαίου και καταπολεμούμε και τα βασανιστήρια και κάθε μορφή καταστολής της ελευθερίας του λόγου. Το νέο ποινικό δίκαιο θα ισχύσει από το Σεπτέμβριο μετά από την αναθεώρηση, όπως προβλέπετε. Έτσι ώστε να συμβαδίσει το λειτουργικό πλαίσιο με την αναθεώρηση του ποινικού δικαίου. Ε, πέρσι γιορτάσαμε την 25η επέτειο της απελευθέρωσής μας και γι' αυτό εγκρίναμε ένα νόμο για την αμνηστία. Όλα αυτά το 2015. Όσοι λοιπόν είχαν ε, εγκληματίσει πριν από το 2014 ή μάλλον μέχρι το 2014 θα απαλλαγούν από τις διαδικασίες δίωξης μέσα στα πλαίσια βεβαίως των ε, αδικημάτων πολιτικού χαρακτήρα, πολιτικών πεπιθήσεων. Άρα το άρθρο 4 ορίζει ότι δεν θα ληφθούν υπόψη αυτά τα δεδομένα και θα δοθεί αμνηστία. Όμως ο Πρόεδρος προέβαλε βέτο σε ορισμένα ε, σημεία του νόμου περί αμνηστίας σε περίπτωση διαφθοράς ε, ε, αντιπίσης αρχής ή ε, περίπτωση κατάχρηση εξουσίας δεν θα ισχύσει αυτός ο νόμος περί αμνηστίας. Έγινε λόγος λοιπόν και συζητήθηκε το θέμα στο Εθνικό μας Κοινοβούλιο και τελικά το Κοινοβούλιο δέχτηκε το βέτο του Προέδρου τον Οκτώβριο το Κοινοβούλιο ενέκρινε ένα νέο νόμο, μία εξαίρεση δηλαδή ως προς την αμνηστία και σαν αποτέλεσμα 1.700 ε, κρατούμενοι απελευθερώθηκαν. Σε αυτή την περίπτωση όταν μιλάμε για διαφθορά ή παράνομη κατοχή κεφαλαίου καθώς και ε, περιπτώσεις ε, κατάχρησης αρχής δεν χορηγήθηκε αμνηστία. Όπως ξέρετε η Μογγολία είναι μέλος του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για την περίοδο 2016-2019. Επειδή έληξε ο χρόνος μου, αργότερα θα απαντήσω σε ερωτήσεις σας. Ευχαριστώ κύριε Πρέσβη. Εσείς τώρα κύριε Λέφλερ της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικών Δράσεων. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, καθώς και την κυρία Συμπρόεδρο. Ευχαριστώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που διεξάγει την παρούσα ακρόαση όπου μας δίνει την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε την κυρία Μάλμστρομ ε, να εξηγεί τι σημαίνει μια πολιτική βασισμένη σε αξίες καθώς και ο συγκερασμός των διαφόρων ε, συμφερόντων που ακούσαμε από τους πρέσβεις των ε, χωρών του Πακιστάν και της Μογγολίας. Είναι σημαντική η συνεισφορά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την εφαρμογή των γενικευμένων προτιμήσεων, ιδίω δε των αντιπροσωπιών του Κοινοβουλίου που προωθούν τα θέματα στις δικαιούχους χώρες και για τις 27 αυτές ε, θεμελιώδεις ε, συνθήκες. Το γενικευμένο σύστημα προτιμήσεων αλλά και το άλλο που λέει οτιδήποτε εκτός όπλων είναι σημαντικά εργαλεία για την ανάπτυξη των αναπτυσσόμενων χωρών. Οι προτιμήσεις GSP μπορούν να συμβάλλουν σημαντικά στην βιώσιμη ανάπτυξη. Ωστόσο, τα ωφελήματα από το σύστημα GSP Plus βελτιώνουν την θέση και των κυβερνήσεων και των εργαζόμενων, ενθαρρύνουν τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις παγκοσμίω να εμπιστεύονται κάποιες ετικέτες ποιότητας και αυτό ισχύει και για τις επενδύσεις. Η συμβολή όλων αυτών στην ε, βιώσιμη ανάπτυξη τονίστηκε και πάλι στο, στα Ηνωμένα Έθνη το Σεπτέμβριο. Μια εμπορική πολιτική βασισμένη σε αξίες συμβαδίζει και με το σχέδιο δράσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα που ε, θα ε, λειτουργήσει μέχρι το 2019 και μέσα στο πλαίσιο του ίδιου στρατηγικού πλαισίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία με πιο στοχευμένη εφαρμογή όλων των εργαλείων αυτών σε όλο το φάσμα. Ένα από τα στοιχεία του νέου σχεδίου δράσεων είναι να περιληφθούν τα στοιχεία αυτά σε όλες τις πολιτικές και δράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο μεταναστευτικό και στην ε, ε, αντιτρομοκρατία και στις επενδύσεις. Εξασφαλίζοντας και προς τα έσω και προς τα έξω συνοχή. Είναι πολύ σημαντικό αυτό στο παρόν πλαίσιο των ε, αυξημένων μεταναστευτικών πιέσεων. Ένα πράγμα το οποίο οφείλω να τονίσω ιδιαίτερα όταν διαβάζω την έκθεση για το GSP είναι ότι δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις για ορισμένες από τις τεράστιες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι χώρες εταίροι μας σε ό,τι αφορά την εφαρμογή των 27 θεμελιωδών συνθήκων. Η εφαρμογή των οποίων συνθήκων σημαίνει αντιμετώπιση σημαντικών προκλήσεων, ιδίως για ε, αυτές τις ευάλωτες αναπτυσσόμενες χώρες. Εκεί μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο οι γενικευμένες προτιμήσεις. Όλες οι χώρες που συμμετέχουν στο σύστημα GSP έχουν κάνει σημαντικές πρόοδους στην εφαρμογή των 27 ε, θεμελιωδών συνθήκων. Όλες έχουν κάνει σημαντικά βήματα και θεσμικά, νομοθετικά και οργανωτικά. Αυτά λοιπόν είναι τα καλά νέα, που όμως δεν αρκούν, διότι αυτό που χρειάζεται εν τέλει είναι η εφαρμογή και η συγκεκριμένη πρόοδος επιτόπου. Όλες οι χώρες αυτές λοιπόν έχουν κάνει βήματα για την εφαρμογή επιτόπου. Καμιά φορά είδαμε πρόοδο, καμιά φορά πολύ περιορισμένη, αλλά θα συνεχίσουμε να ασκούμε πίεση ώστε να σημειωθεί και άλλη πρόοδος. Ε, αυτό θα πρέπει να είναι και στο επίκεντρο της προσπάθειας monitoring της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κύριε Συμπρόεδρε, αυτό το monitoring έχει δώσει και άλλες αφορμές και ευκαιρίες για να εφαρμοστούν ε, τα συστήματα των γενικευμένων προτιμήσεων με ναι, ενίσχυση του διαλόγου για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα δικαιώματα των εργαζόμενων, την ε, αηφόρο ανάπτυξη και την χρηστή διαχείριση. Παράδειγμα το Περού, όπου έχουν σημειωθεί σημαντικές πρόοδοι. Το ίδιο για την περίπτωση της Μογγολίας που ακούσαμε λίγο πριν. Αρχίζει και ο πρώτος διάλογος ανθρώπινων δικαιωμάτων μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Μογγολίας αργότερα, φέτο θα γίνουν και ε, αποστολές monitoring στην Βολιβία και στην Παραγουάη για θέματα που θα καλύψουν ζητήματα ανθρώπινων δικαιωμάτων. Η Επίτροπος Μάλμστρομ έδωσε ορισμένα παραδείγματα σχετικά με το τι πράττουμε και πώς αξιολογούμε τις ε, εξελίξεις στην Μογγολία και στην Αρμενία. Εγώ θα ήθελα να προσθέσω εδώ λίγα λόγια για το Πακιστάν. Στα συμπεράσματα το έγγραφο λέει οι παραβιάσεις ανθρώπινων δικαιωμάτων εξακολουθούν να είναι εκτεταμένες στην χώρα αυτή παρόλες τις σημαντικές επικοδομητικές προσπάθειες. Έχει επιτευχθεί πρόοδος στην ενίσχυση του θεσμικού πλαισίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Έχει μάλιστα ιδρυθεί και Εθνική Επιτροπή Ανθρώπινων Δικαιωμάτων καθώς και άλλοι θεσμοί και Επιτροπή Εφαρμογής του συστήματος GSP που εκπροσωπεί σήμερα εδώ ο κύριος Άλλη και δια του προσώπου του επιθυμώ να συγχαρώ την πακιστανική κυβέρνηση για τις προσπάθειες της αυτές. Σημαντικές είναι και προσπάθειες του Ανωτάτου Δικαστηρίου για την εξασφάλιση της ανεξαρτησίας του ρόλου του καθώς και για την ενημέρωση και ο ρόλος που παίζει η κοινωνία των πολιτών για την προσέγγιση των ανθρώπινων δικαιωμάτων και στην χώρα αυτή αλλά και διεθνώς. Το, Πακιστάν έχει υποβάλει και σχετικές εκθέσεις. Τι κάνουμε τώρα για να ενισχύσουμε τις προσπάθειες αυτές των χωρών GSP+, εκτός από το διάλογο. Με το Ευρωπαϊκό Εργαλείο για τη Δημοκρατία και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε να υποβληθούν προτάσεις για τη συνεργασία με τους ε, εταίρους για την εφαρμογή της νομοθεσίας GSP. Αυτό έγινε το 2015. Θα επιλεγούν έργα, project δηλαδή, σχέδια, στην διάρκεια του 2016. Τα project που θα επιλεχθούν θα αρχίσουν να εφαρμόζονται στο τέταρτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους. Και αυτό αφορά έξι από τις χώρες αυτές για την εφαρμογή 8 συνθήκων του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας. Κύριε Συμπρόεδρε, το σύστημα GSP Plus αποτελεί και μια γέφυρα για την ενισχυμένη συνεργασία των κεφαλαίων βιώσιμης ανάπτυξης για τις ε, συμφωνίες ελευθέρων συναλλαγών. Πολλά μείνουν να γίνουν ακόμη, ιδίως σε ό,τι αφορά τις υποεπιτροπές εμπορίου και ε, αηφόρου ανάπτυξης. Αυτά που έμαθαν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η υπηρεσία μας είναι δεν υπάρχει το one size fits all. Για παράδειγμα, το πράσινο ακροτήρι, κάπε βέρντε. Χώρα η οποία δεσπόζει στην περιοχή της λόγω του καλού της ιστορικού προστασίας ανθρώπινων δικαιωμάτων. Και ωστόσο έχει προβλήματα. Το Πακιστάν, το οποίο αντιμετωπίζει τεράστια προβλήματα ασφάλειας. Και μια χώρα όμως η οποία εγκύπτει σοβαρά στην προσπάθεια με την λήψη θεσμικών μέτρων. Στη βάση των εμπειριών αυτών θα εκδώσουμε τώρα κατευθυντήριες γραμμές για την επόμενη περίοδο monitoring ώστε να ενστερνιστούν οι ε, χώρες αυτές να αναλάβουν την διοκτησία δηλαδή των μεταρρυθμίσεων αυτών. Η Κομισιόν και η Υπηρεσία μας Εξωτερικών Δράσεων θα προχωρήσουμε στη συνεργασία με τις ε, δικαιούχους χώρες και σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο Πρόεδρος. Σας ευχαριστώ πολύ. Έχουμε λοιπόν τώρα ακριβώς 15 λεπτά στη διάθεσή μας για να θέσουμε ερωτήσεις. Υπενθυμίζω ότι πρόκειται για ερωτήσεις. Μην προβείτε σε τοποθετήσεις. Να ρωτήσετε, να απευθύνετε ερωτήσεις στους ειδήμονες μπορώ να διαθέσω 2,5 λεπτά για κάθε, ε, συγγνώμη, 1,5 λεπτό για κάθε ερώτηση. 1,5 λεπτό για κάθε ερώτηση. Πρώτα ο εισηγητής και σκιώδης εισηγητής για 1,5 λεπτό όπως είπα. Ευχαριστώ Πρόεδρε, πολύ σύντομα. Το σύστημα GSP Sin περιλαμβάνει ήδη κάμποσες χώρες που συμμετέχουν αλλά εποφελούνται και άλλες χώρες μέχρι τη λήξη του συστήματος το 2023. Θα πρέπει λοιπόν, εάν αποφασίσουμε κάτι γι' αυτό, να αποφασίσουμε καιρό στην παράτασή του. Πάντως υπάρχουν χώρες που μπορούν να αφήσουν το σύστημα αυτό, είτε παίρνοντας ε, ένα πτυχίο, για να το πω έτσι, γινόμενες χώρες μέσω εισοδήματος, είτε συνάπτοντας μια συμφωνία ελεύθερου εμπορίου. Αυτή είναι και η αξία του συστήματος. Αυτό που θα ήθελα λοιπόν να ακούσω από τις χώρες και τους εκπροσώπους τους που έχουμε εδώ, είναι πώς ε, οι οικονομικές τους επιδόσεις έχουν αλλάξει. Πόσο περιμένουν να χρειαστούν παραμονή στο σύστημα. Τι ε, πιστεύουν οι ίδιοι. Γιατί φαντάζομαι θα τους έχει απασχολήσει. Ευχαριστώ. Η κυρία Μόσκα. Ευχαριστώ πρόεδρε. Μια πολύ συγκεκριμένη ερώτηση. Οι βελτιώσεις από την πλευρά της πακιστανικής κυβέρνησης. Ακούσαμε πως υπάρχει προσαρμογή βάσει των προκρατήσεων του συστήματος GSP-SYN ιδίως στους τελευταίους μήνες και ξέρουμε τι ισχύει για τον τομέα των κλωστιοϊφαντουργικών. Ξέρουμε ότι στον τομέα αυτό υπάρχει μεγάλη γυναικεία παρουσία μεταξύ του εργατικού δυναμικού. Η κατάσταση όμως των γυναικών στο Πακιστάν δεν έχει βελτιωθεί συγκριτικά σε σχέση με τον όγκο των εξαγωγών που αυξήθηκαν. Αυτή είναι μια συγκεκριμένη περίπτωση. Μας επιτρέπει να κοιτάξουμε πώς πέραν του ελέγχου και της εποπτείας που είναι πολύ σαφής, μπορεί κανείς να παρέμβει για να βελτιώσει την δράση μας, τη δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε στην ε, χώρα να υπάρχει πιο αποτελεσματική εφαρμογή και να δώσει ε, ωφέλη ισορροπημένα και στο επίπεδο των δικαιωμάτων όπως και των οικονομικών ωφελών. Για τα δικαιώματα των γυναικών ξέρουμε πως ε, στον τομέα αυτό δεν υπάρχει απαραίτητη δράση, απαραίτητη παρέμβαση από τις κεντρικές αρχές. Καρίμ. Ευχαριστούμε. Καρίμ. Ευχαριστώ Πρόεδρε, Συμπρόεδρε, Επίτροπε. Να ξεκινήσω λέγοντας ότι έχω άμεση εμπειρία από το πόσο επιτυχημένο είναι το πρόγραμμα αυτό ώστε η Ευρώπη να αναλαμβάνει υποχρεώσεις και να τις εκπληρώνει. Είχαμε υποψίες από το σώμα κάποιες φορές ότι ήταν ένα, μια θεσμική ε, το σύστημα αυτό. Όμως ακούω τις δεσμεύσεις και της ε, Επιτρόπου Μαλστρόμ και ξέρω και πόσο ο συνάδελφος Φιέλνερ προωθεί τα θέματα αυτά, οπότε ξέρω ότι όλοι δεύουμε προς την ίδια κατεύθυνση. Κυρία Μαλστρόμ, δύο θέματα θέλω να θέσω για την διαφοροποίηση. Ένας από τους βασικούς στόχους όσων προσπαθούμε να κάνουμε είναι ότι θα διευρύνουμε και θα ενδυναμώσουμε τις οικονομίες με τις οποίες ξεκινούμε να έχουμε σχέσεις. Έχω συγκεκριμένες ευθύνε για την Αρμενία, τη Γεωργία και ad hoc για το Πακιστάν επίσης. Δεν βλέπω να υπάρχει απαραίτητη μόχλευση για να ενθαρρύνουμε την διαφοροποίηση. Κατά δεύτερον, ως προς το πώς θα προχωρήσουμε στο επόμενο βήμα ή ακόμη παραπέρα. Έχω την αίσθηση ότι ο συσχετισμός ε, εταιρείε προς εταιρείε, B2B από ευρωπαϊκές προς τις εταιρείε του Πακιστάν ή της Αρμενίας δεν προχωρούν αρκετά. Έχει σκεφτεί η Επιτροπή να θεσπίσει προγράμματα για να προωθήσει αυτού την ανάπτυξη. Πρόεδρε, την επόμενη φορά μου χρωστάτε 7 δευτερόλεπτα. Εντάξει λοιπόν. Ο κύριος Σόλτ. Σας ευχαριστώ. Και εγώ θα ήθελα να είμαι συνοπτικός. Σας ευχαριστώ για τις ενημερώσεις και τις παρουσιάσεις Έχω δύο ερωτήσεις προς την Επίτροπο Μάλστρομ και στον πρέσβη του Πακιστάν. Ακούσαμε ότι η πακιστανική κυβέρνηση και ο πρέσβης ερμηνεύουν την κατάσταση ως βελτιωμένη ως προς το πώς ε, προστατεύονται τα ανθρώπινα δικαιώματα συγκεκριμένα. Αλλά έχουμε και ειδήσει και νέα, καθώ και αυτόπτες μάρτυρες, ότι η κατάσταση δεν είναι και τόσο καλή τόπου όπως συχνά περιγράφεται εκτό. Ποια είναι λοιπόν η θέση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή τώρα να ακούγονται αυτέ οι κρίσει για την βελτίωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και εμεί μπορεί να ακούμε ότι υπάρχουν παραβιάσει. Υπάρχει τέτοιο κριτήριο για το καθεστώ GSP και gsp μπορούμε να αποτιμήσουμε κάποια στιγμή αν πραγματικά λειτουργούν τα εργαλεία μας. Και έχω επίσης και την προτροπή προς την Πακιστανική κυβέρνηση και τον πρέσβη, αλλά και ερώτηση. Πώς ερμηνεύετε εσείς εντός της χώρας σας αυτές τις ε, ενδείξεις. Πολλές από τι εξελίξεις στη χώρα σας δεν είναι τόσο ικανοποιητικέ. Πώς θέλετε να ξεπεράσετε τα προβλήματα, να καλύψετε τα χάσματα στην κοινωνία σας. Πώς καταγράφετε το που έχετε φτάσει στο να αντιμετωπίσετε και να καλύψετε τις προσδοκίες του Ευρωκοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα πλαίσια του καθεστώτος συν Ευχαριστούμε, κύριος Βόχνερ. Επίτροπε Μάλστρο, μιλήσατε για πρόοδο στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Όμως, υπάρχουν και σοβαρές οπισθοδρομήσεις. Εδώ μιλάω για την άρση του μορατόριου για τη θανατική ποινή στο Πακιστάν, που δεν οδήγησε σε καμία αντίδραση από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ε, πέραν από δύο γραμμές έκφρασης δυσαρέσκειας σε μια έκθεση 308 σελίδων. Το Συμβούλιο ξεκάθαρα θέλει το Πακιστάν ε, στη συνεργασία του και στο συμπεράσματα του Ιουλίου 2015 αναφέρεται ότι η άρση του μορατόριου για τη θανατική καταδίκη αντιφάσκει με το καθεστώς GSP-SYN εσείς τι κάνετε, απλώς αγνοείτε την τοποθέτηση του Συμβουλίου και έχω μια δεύτερη σημαντική ερώτηση. Ένας ευρύς συνασπισμό με κυβερνητικών οργανώσεων ζητά ανεξάρτητη επισκόπ, ε, έρευνα για την ε, θανατική καταδίκη και την επανεισαγωγή άλλου μορατόριου βάσει των αποτελεσμάτων της έρευνας που θα γίνει θα μπορούσε η DigiTrade να τρέξει στο άρθρο 15 της συνθήκης για να αποκλείσει τελείως το Πακιστάν από το καθεστώς GSPC. Εσείς απαντήσατε στον συνασπισμό των μη κυβερνητικών οργανώσεων για το θέμα αυτό και θα μπορούσατε να μας πείτε εδώ στους ευρωβουλευτές την άποψή σας για αυτό το θέμα. Ευχαριστώ. Ο κύριος Φαντάλεν. Θα μιλήσω Ολλανδικά, οπότε ίσως να χρειαστείτε τα ακουστικά σας. Έχω μια ερώτηση για την Επίτροπο. Για το Πακιστάν. Όταν ε, συμμετείχαμε, αρχίσαμε να συμμετέχουμε στο σύστημα GSP SYN, ήδη δεν σεβόταν τα ανθρώπινα δικαιώματα του Πακιστάν και αυτό εξακολουθεί. Η κυβέρνηση διαρκώ παραβιάζει τα δικαιώματα των πολιτών. Ο ΙΕ λέει ότι όσα γίνονται εκεί δεν συνάδουν με τη σύμβαση. Εσείς λέτε ότι το Πακιστάν χρησιμοποιεί τη θανατική καταδίκη για πολύ σοβαρά εγκλήματα μόνο. Και ότι μόνο τότε εφαρμόζεται η θανατική ποινή. Αυτό όμω στην πραγματικότητα δεν φαίνεται να ισχύει. Το Πακιστάν δεν εκπληρώνει μια σειρά από τι υποχρεώσει του βάσει των διεθνών ε, συμφωνιών και των θεμελιωδών συμβάσεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τι θεμελιώδει ελευκαιρίε. Πώ γίνεται λοιπόν παρά την κατάσταση αυτή να μην λαμβάνετε μέτρα κατά το Πακιστάν. Δεν καταλαβαίνω τι δηλώσει σα. αυτές οι συμβάσεις δεν γίνονται σεβαστές και δεν αναλαμβάνεται δράση. Θα ήθελα να πω το εξής προς την Επίτροπο. Χαίρομαι διότι εφαρμόζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα σε παγκόσμιο επίπεδο και ξέρω ότι η κατάσταση στο Πακιστάν είναι πολύ λεπτή εξαιτίας των τρομοκρατικών ε, δραστηριοτήτων. Αλλά όπως ξέρετε υπήρξε μορατόριου ως προς τη θανατική ποινή και όπως ξέρετε πρόκειται να εκτελεστούν άμεσα 113 άνθρωποι. Αυτοί που επίκειται να εκτελεστούν είναι μεταξύ των 1.000 και των 1.500. Νομίζω ότι θα πρέπει στο Πακιστάν να ε, αναθεωρηθεί ο ποινικό κώδικας και να δούμε πώς, ε, ποια είναι η κατάσταση αυτών των ανθρώπων. Θα ήθελα να μου πείτε πώς ε. έχει το ζήτημα και πώς είναι η κατάσταση και ποια μέτρα θα λάβει η κυβέρνηση του, του Πακιστάν επί του θέματος. Κύριε Ροντρίγκε, ευχαριστώ Πρόεδρε. Εντάχει θα ήθελα να ευχαριστήσω του πρέσβης του Πακιστάν και της ε, Μογγολίας που παρευρίσκονται και την Επίτροπο ε, Μάλμστρεμ. Σε σχέση με αυτά που είπε ο κύριος Φίσας, γνωρίζουμε τις δυσκολίες ε, του Πακιστάν να αντιμετωπίσει την τρομοκρατία, αλλά είναι γεγονός ότι το 2008 εισήχθη αυτό το μορατόριουμ για την θανατική ποινή και ο πρόεδρος Σαρίφ δυστυχώς ε, τη, το επανεισήγαγε. Η μεγάλη σφαγή στο κολέγιο εκείνο του Πακιστάν μας ε, δείχνει, στο σχολείο του Πακιστάν, δείχνει πώς έχει κατάσταση. Όπως ξέρετε ε, αυτή τη στιγμή επίκειται η θανατική ποινή για 300 ε, περίπου ανθρώπους. Πέρα από την πρόοδο που έχει γίνει στο Πακιστάν ε, για, ως προς τα ανθρώπινα δικαιώματα, θα ληφθεί υπόψη το αίτημα του, των Ηνωμένων Εθνών σε σχέση με το, την άρση του μορατόριου και να μην γίνονται εκτελέσεις ανηλίκων κυρίως. Θα ήθελα να μου πείτε πώς ε, μπορούμε να βοηθήσουμε εμείς έτσι ώστε να προωθηθούν ε, τα ανθρώπινα δικαιώματα πληρέστερα σε αυτές τις χώρες. Ευχαριστώ. Εγώ είμαι μέλος της Υποεπιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και θα ήθελα να σταθώ σε αυτό που είπε και η Αντιπρόεδρός μας, δηλαδή πώς θα, ε, συμμετάχει, θα μας συμμετάσχει η κοινωνία των πολιτών στην όλη διαδικασία αυτή. Η ερώτηση είναι προς εσάς και προς τον κύριο Λέφλερ. Στην ε, ε, διαδικασία αναθεώρησης του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών υπάρχει ένας μηχανισμός προόδου έτσι ώστε να συμμετέχει γενικότερα και η κοινωνία των πολιτών σε αυτά τα, τα δρόμενα. Θεωρείτε ότι μπορεί να υπάρξει έλεγχος και στα πλαίσια του GSP Plus και σε τοπικό και σε εθνικό επίπεδο. Πισέρα. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να σταθώ στα ερωτήματα των συναδέλφων σε σχέση με την εξέλιξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Πακιστάν και ιδιαίτερα τη θανατική ποινή. Νομίζω ότι μιλάμε για βελτίωση των, της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και αυτή η αναθεώρηση και θα ήθελα να ρωτήσω ποια είναι τα σχέδια της κυβέρνησης έτσι ώστε κατά την προσεχή αναθεώρηση να μην έχουν ε, ήδη θανατωθεί χίλιοι άνθρωποι. Θα ήθελα να μου πει η Επιτροπή ποιους μηχανισμούς προβλέπει μια διερευνητική διαδικασία ή κάτι έναντι του ε, Πακιστάν. Και θα ήθελα να πω ότι χαίρομαι που έχει καταργηθεί η παιδική εργασία. Ως προς τη Μογγολία θα ήθελα να ρωτήσω, στο νέο ποινικό κώδικα θα ε, γίνει λόγος για την ε, απαλυφή των βασανιστήριων. Ο κύριος Λέφλερ μίλησε για, και, για το, και άλλα θέματα. Εμείς στην ε, Υποεπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ασχοληθήκαμε και με το θέμα της Γουατεμάλας και τις ε, γενικευμένες προτιμήσεις ιδιαίτερα ως προς τις, ε, τη διάκριση κατά των γυναικών και των παιδιών. Ε, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους ομιλητές. Χαιρόμαστε, χαίρομαι γιατί μιλάμε για τις θετικές εμπειρίες όπου υπάρχει καλύτερος διάλογος, καλύτερη μόχλευση για να φτάσουμε σε καλύτερα αποτελέσματα. Επίτροπε, αναφερθήκατε στο γεγονός ότι η Επιτροπή θα ήθελε να αναστείλει τις γενικευμένες προτιμήσεις αν αυτό πρέπει να γίνει και όπου πρέπει να γίνει. Ποια είναι τα κριτήρια που θα ακολουθηθούν γιατί στη Γουατεμάλα ακόμα κι αν υπάρχουν ε, δύο παράγραφοι του ILO που δείχνουν ότι γίνεται συστηματική παραβίαση των βασικών συμβάσεων και μέσα στα πλαίσια του GSP+, δεν είδαμε κάποια δράση από την Επίτροπη. Επίσης, σε σχέση με τις ε, κατεξιότηση πράξης για την συστηματική μη εφαρμογή συμβάσεων, θα πρέπει να ορίσουμε ένα κατόφλι, κάτι το οποίο δεν είδαμε τα τελευταία δύο χρόνια. Δεσμεύεστε να υπάρξει μια κατεξουσιοδότηση πράξη, γιατί έτσι θα υπήρχε διαφάνεια για το πώς ε, εφαρμόζονται αυτά τα κριτήρια από πλευράς ε, της Κομισιόν. Έχω μια πολύ απλή ερώτηση για την Επιτροπό και δεν θα χρειαστώ όλο το χρόνο μου. Αλλά σε άλλη ευκαιρία, αν παραδειγματιστώ από τον συνάδελφο, θα, μένα, θα μου χρωστάτε ένα λεπτό, Πρόεδρε. Για το σύστημα GSP GSP-SYN και κατά την άποψη τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο πρωταρχικό σκοπό του συστήματο ποιο είναι, να βοηθήσει τι αναπτυσσόμενε χώρε, ή ο πρωταρχικό σκοπό του συστήματο αυτού είναι να προωθήσει την πολιτική ατζέντα και τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ελπίζω να μην αποφύγετε να απαντήσετε στην ερώτηση όταν δώσετε απαντήσεις. Από την Ινδονησία, από το Steering Committee, ένας ε, συνάδελφος μας ζήτησε το λόγο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η Ινδονησία είναι μία από τις χώρες που επωφελούνται από το σύστημα GSP+. Θα ήθελα να έχω κάπως περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το εξής. Πώς εφαρμόζει το σύστημα GSP συν η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ποιος είναι ο ρόλος του Κοινοβουλίου σας στο σύστημα αυτό και πώς παρακολουθείτε την εξέλιξη του συστήματος. Για ορισμένα προϊόντα, όπως, αχαρο, όπως για το κρέας τόνου σε κονσέρβες, αλλά και για τους ανανάδες σε ε, κονσέρβες, εποφελούνται από το GSP-SYN πώς παρακολουθείτε τα ανθρώπινα δικαιώματα σε τέτοιες χώρες. Από την 1η Ιανουαρίου του 2015, 2014 ε, με συγχωρείτε, ορισμένες κατηγορίες προϊόντων έχουν αποκλειστεί αφορώντας χώρες όπως Κίνα, Ινδία, ε, Ουκρανία και Νιγηρία. Η Ινδονησία ε, εποφελείται εκτός από ζωντανά ζώα φυτικά η ζωικά έλαια, χημικές ουσίες άλλες εκτός από οργανικές. Η ερώτησή μου λοιπόν είναι η... πώς παρακολουθείτε τις χώρες που δεν επωφελούνται πλέον από τις ε, προτιμήσεις. Τώρα, έχω και εγώ δύο ερωτήσεις. Πρώτα και την κυρία Μάμψον και τον κύριο Λέφλερ. Το ερώτημα είναι, αυτές οι 27 θεμελιώδεις συνθήκες που οφείλουν να τηρούνται. Αυτό είναι σημαντική πρόκληση. Δεν χρειαζόμαστε λοιπόν ένα ξεκάθαρο δικό χάρτη με ορόσημα πότε πρέπει να εφαρμοστεί ποιο πράγμα. Δεύτερο, ο μηχανισμός εμπλοκής της κοινωνίας των πολιτών. Πώς εξασφαλίζεται. Δεν θα ήταν σωστό αναέτος να οργανώνεται στρογγυλή τράπεζα με οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών για να υπάρχουν και ανεξάρτητες γνωμοδοτήσεις σχετικά με την εφαρμογή των συνθήκων αυτών. Και το μοντέλο των πακιστανικών συνδικάτων, δηλαδή αν ε, υποβολή ανεξάρτητης έκθεσης, δεν θα μπορούσε να αποτελέσει πρότυπο και για άλλες χώρες για να έχουμε μια βασική εικόνα σχετικά με την εφαρμογή των ε, συνθήκων αυτών. Και τρίτο, κυρία Μάλμστρομ, σχετικά με την διαδικασία αναθεωρήσεως. Μας μένουν 8 χρόνια μέχρι να συμπληρωθεί ο ορίζοντας των 10 ετών και θα χρειαστούμε μετά βεβαίως ένα διάδοχο του συστήματος GSP. Θα δώσω το λόγο τώρα στους ειδήμονες και πρώτα στην κυρία Μάλμστρομ. Μάλιστα, ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω να απαντήσω στις ερωτήσεις, ορισμένες επικαλύπτονταν βέβαια και ξεκινώντας από το Πακιστάν. Αν ε, διαβάσετε την έκθεση στο σύνολό της, μόνο 350 σελίδες είναι, πιστεύω θα τα έχετε διαβάσει όλοι, θα είδατε, όπως είπε και η κυρία Κίτον Ντάρλινγκ, ότι τονίζουμε τα Είναι σημαντικό να πει κανείς ότι όλες αυτές οι χώρες καταβάλουν προσπάθεια. Όλες αυτές οι χώρες δημιουργούν θεσμούς και είναι πολύ επικοδομητικός ο διάλογος μαζί τους και βλέπετε συγκεκριμένα βήματα πρόοδου. Όμως πολλές χώρες έχουν ακόμα σημαντικά προβλήματα ανθρώπινων δικαιωμάτων. Σημαντικά προβλήματα σε ό,τι αφορά το, την δυνατότητα να αρθούν στο ύψος του επίπεδου των διεθνών συνθήκων. Η κατάρριση της ποινής ε, υπό αυστηρούς όρους δεν είναι δεν ε, περιλαμβάνεται σε μία από τις 27 αυτές συνθήκες. Εγώ έχω μιλήσει με τον Υπουργό κατ' επανάληψη για την κατάργηση του μορατόριου. Μας απασχολεί αυτό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πιέζει διαρκώς για την κατάργηση της θανατική ποινής. Όμως Υπό αυστηρή έννοια δεν είναι στο περιεχόμενο κάποιες από τις 27 συνθήκες. Παρ' όλα αυτά συνεχίζουμε να, ασκήσουμε, να ασκούμε πίεση. Πώς παρακολουθούμε, πώς κάνουμε το monitoring. Συνεργαζόμαστε ιδίω όσοι γνωρίζετε με τα Ηνωμένα Έθνη και τον Διεθνή Οργανισμό Εργασίας και με τις ε, ε, οργανώσεις κοινωνίας των πολιτών μέσω των αντιπροσωπιών μας. Θα συζητήσω μαζί σας εάν μπορούμε ενδεχομένως να εντείνουμε τον διάλογο με πιο συστηματικό τρόπο. Σε ορισμένες χώρες μέλη υπάρχει μια πολύ έντονα κινητική κοινωνία των πολιτών, αλλού όχι. Γι' αυτό συνεργαζόμαστε και με τα Ηνωμένα Έθνη και με τον ILO που έχουν μεγάλη εμπειρία. Βεβαίω και εγώ, αλλά και άλλοι, βρισκόμαστε σε διαρκή επαφή με οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και τα θέματα αυτά επανέρχονται διαρκώς. Είναι πολύ δύσκολο να υπάρξουν κατεξουσιοδότηση πράξεις για την αντιμετώπιση σοβαρών παραβιάσεων. Βεβαίως εντοπίζονται διαρκώς διαφορετικά τέτοια θέματα. Αυτό που προσπαθεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι να θεσπίσει ένα διάλογο και να δει αν αυτός μπορεί να αποδώσει. Εάν επιλέξει βέβαια στον επόμενο γύρο εποπτείας, αν καταρρίξει μάλλον, ότι υπάρχουν βήματα οπισθοδρομήσεως, τότε θα αποσύρουμε τις γενικευμένες προτιμήσεις από τη συγκεκριμένη χώρα. Αυτό όμως θα έχει και σημαντικές επιπτώσεις και στην κοινωνία των πολιτών. Μπορεί να έχει κάποιο συμβολικό αποτέλεσμα. Μπορεί να, είναι σημαντικό. Ή μπορεί να χρειαστεί να προσφύγουμε σε άλλες μορφές διαλόγου που να αποφέρει καλύτερα αποτέλεσματα. Συνεργασία λοιπόν με τον ΑΕΛΟ, με τα Ηνωμένα ΕΕ, Έθνη, με τι κυβερνήσει και σε ελληνικές περιπτώσει και με οργανώσει τη κοινωνία των πολιτών. Είναι πολύ δύσκολο λοιπόν αυτό. Γι' αυτό και αυτό το engagement, η εμπλοκή είναι το πιο σημαντικό, η πιο σημαντική προσπάθεια. Σε ό,τι αφορά το Πακιστάν, κυρία Μόσκα, η κατάσταση των γυναικών είναι εκεί ε, από τις προτεραιότητές μας. Βεβαίως, θεσπίστηκε εντωμεταξύ κάποια ε, νομοθεσία με θετικό πρόσημο για τις γυναίκες. Είναι πολύ σημαντικό, αλλά χρειάζεται να συνεχιστεί η προσπάθεια. Αγαπητέ μου, Κόμι, Ποτέ δεν αποφεύγω τις ερωτήσεις σας. Ο στόχος μας είναι να βοηθήσουμε τις χώρες αυτές. Πρωτίστως. Αυτός είναι ο πρωταρχικός μας στόχος. Πώς θα το κάνουμε αυτό. Τις βοηθούμε ανοίγοντας τις αγορές μας. Έτσι ώστε να αυξηθούν οι εμπορευματικές ροές και να δημιουργηθούν περισσότερες δυνατότητες υπέρ των ανθρώπων αυτών. Διαδίδουμε τις αξίες μας, ναι, αλλά είναι παγκόσμιες αξίες. Γι' αυτό είπαμε ότι αυτές οι 27 θεμελιώδεις διεθνείς συνθήκες, δεν είναι ευρωπαϊκές συνθήκες αυτές, είναι το κλειδί για να υπάρξει πρόσβαση στο σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων. Υποστηρίζουμε τις χώρες αυτές λοιπόν έτσι ώστε να βελτιώσουν τη δημοκρατία τους, τις δυνατότητες για τους πολίτες τους και ταυτόχρονα προωθούμε ευρωπαϊκές και διεθνές αξίες. Αυτά, κύριε Πρόεδρε, νομίζω απήντησα. Υπάρχουν και άλλοι βεβαίως που μπορούν να συμπληρώσουν. Η θανατική ποινή. Όπως είπα προηγουμένως, χάθηκαν ζωές τόσων αθώων, 60.000 άμαχοι, που θανατώθηκαν, παιδιά θανατώθηκαν. Γιατί γιατί τους εκδικήθηκαν. Τα φέρετρά τους ήταν αδύνατο να τα βαστάξει κανείς. Και το λέω αυτό πραγματικά με βαριά καρδιά. Είμαστε όμως σε κατάσταση πολέμου. Είναι ένας πόλεμος που συνεχίζεται αμύωτος. Βρισκόμαστε σε μια κατάσταση όπου είμαστε τρομοκρατημένοι. η Επιτροπή σας και το έξοχο ε, σώμα σας εύχομαι να δείτε τα πράγματα από αυτή την προοπτική. Δείτε το θέμα και έτσι. Δεν είναι κανονική ποινή ή θεματική. Υπάρχουν πολλές διαβαθμίσεις. Μίλησα για το πρόγραμμα δράσης προηγουμένως. Αυτό το επινοήσαμε για να ξαναδούμε όλους αυτούς τους νόμους, τον ποινικό μας κώδικα ολόκληρο και άλλους ποινικού νόμους που χρήζουν ιδιαίτερη προσοχή. Η πρόοδος είναι υπαρκτή, ίσως να είναι αργή, αλλά είναι βεβαία. Υπάρχει και θα τηρώ ενήμερη την Επιτροπή σα για το τι πρόοδο πραγματοποιούμε. Το Εθνικό Πρόγραμμα Δράσης είναι βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Τα δικαιώματα των γυναικών. Νομίζω ότι έχουμε την πρωτιά ως Πακιστάν να έχουμε τέσσερις γυναίκες πρέσβυρες σε κέρυες θέσεις, εδώ, στη Γενέβη, στη Νέα Υόρκη, και στην Αυστρία. Την τελευταία χρονιά είχαμε τον υψηλότερο αριθμό κυριών στο διπλωματικό δυναμικό αλλά και στα κλωστιντεφαντουργικά και από τις δημόσιες υπηρεσίες έχουμε το μεγαλύτερο αριθμό γυναικών γιατρών. Και αν χρειαστεί μπορώ να σας δώσω και τους ακριβείς αριθμούς. Έχουμε σχετική νομοθεσία, πολύ σοβαρή νομοθεσία, για την εξάλληψη της διακριτικής μεταχείρισης. Και για να προστατευτούν οι κυρίες που εργάζονται σε όλους τους τομείς, τον ιδιωτικό, και έχουμε και ειδικού διαμεσολαβητές και διαμεσολαβήτριες που εξετάζουν αυτά τα τομέα και τα, θέματα και επιβλέπουν αυτούς τους τομείς. Και μην ξεχνάμε Εάν σκεφτόμαστε λίγο εκτός της παπατημένης οδού, εκτός των όσων θα μας έλεγαν οι επιστήμονες και οι καθημαϊκοί, θα ήταν ο κόσμος μας ένα πιο ωραίο μέρος για να ζει κανείς στο μέλλον. Ευχαριστούμε ο πρέσβης από την Μογγολία. Θα ήθελα να προσθέσει κάτι. σε σχέση με το νέο ποινικό κώδικα τον οποίο εγκρίναμε το προηγούμενο Σεπτέμβριο αυτοί που έλαβαν τις αποφάσεις τόνισαν ότι πρόκειται για συνεργασία πολλών ε, ειδημόνων και εμπειρογνωμόνων, επιστημόνων και ούτω καθεξής ε, από το εθνικό και διεθνές στερέωμα για να αλλάξει η κατάσταση στη Μογγολία και ο νέος ποινικό κώδικας αποτελεί κάτι το καινοτόμο και εστιάσε την προσοχή σε, στα βασανιστήρια, στην κράτηση, στις κρατήσεις, στις συλλήψεις και ούτω καθεξής. Αυτοί οι μηχανισμοί θα πρέπει να αλλάξουν. Θα πρέπει να αρθούμε στα διεθνή πρότυπα χρησιμοποιώντας τις νέες τεχνολογίες εποπτείας και παρακολούθησης, καλύτερες συνθήκες ε, κράτησης για τους κρατούμενους και τήρηση των, ε, των ποινών. Και βεβαίως ε, εξέβρεση και άλλων μέσων εναλλακτικών της κράτησης. Επίσης, ο νέος ποινικό κώδικας προβλέπει ότι όλες οι νομικές πράξεις που αφορούν την εφαρμογή του ποινικού κώδικα θα αναθεωρηθούν για να επιλύσουμε και το θέμα των βασανιστήριων. Λέφλερ. Για, να συμπληρώσω αυτά που είπαν οι άλλοι ομιλητές και ιδιαίτερα η Αντιπρόεδρος Μάλμστρομ, η κυρία Λόχ Μπίλερ μίλησε για το ρόλο της κοινωνίας των πολιτών. Με βάση την εμπειρία μου ε, στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών, όπως είπα εξ αρχής, ένα από τα βασικά στοιχεία στην εργασία μας για να εφαρμόσουμε το GSP Plus είναι να έχουμε μια κοινή προσέγγιση για τις γενικευμένες προτιμήσεις, για το πώς δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση προωθεί τις σχέσεις με τις χώρες εταίρους, προωθώντας αυτό τον διάλογο Είπατε ότι θα πρέπει να μη σκεφτόμαστε με βάση μία προδιαγεγραμμένη πορεία. Αυτό είπε ο Πακιστανός πρέσβης. Δηλαδή, να σκεφτόμαστε εκτός πεπατημένης. Και αυτό κάνουμε βαθμία. Το κάνουμε σε ολοένα και περισσότερες χώρες μέσα στα πλαίσια του συστήματος γενικευμένων προτιμήσεων Plus. Συνεργαζόμαστε με το Διεθνή Οργανισμό Εργασίας για να δούμε πώς αποτιμά την κατάσταση. Συνεργαζόμαστε με κυβερνήσεις μέσω διαλόγου και όπως είπε και ο κύριος Άλλη, μιλάμε για τους νέους φορείς και αυτό το κάνουμε βαθμιαία για να ε, μπορέσουμε να έχουμε έναν διάλογο με τη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών για πρώτη φορά και στη Μογγολία. Αυτό το καταφέραμε και με το Περού. Δηλαδή μιλάμε για τα ανθρώπινα δικαιώματα με τη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών. Αυτό αφορά και άλλες χώρες της Λατινικής Αμερικής. Πιστεύω ότι θα πρέπει να συμμετέχει η κοινωνία των πολιτών στην τήρηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και αυτό ισχύει και σε άλλες χώρες της Λατινικής Αμερικής όπως τη Γουατεμάλα. Τώρα, τι κάνουμε ως προς τη Γουατεμάλα και σε σχέση με την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης προσπαθούμε να το προωθήσουμε αυτό το θέμα Μιλάμε για τα δικαιώματα των εργαζομένων, των γυναικών και ούτω καθεξής που είναι αναπόσπαστο τμήμα της ατζέντα με τη Γουατεμάλα. Ως προς τις συμβάσεις ε, του ΔΟΕ συνεργαζόμαστε με τη Γουατεμάλα και δεν ξέρουμε κατά πόσο θα πρέπει να συσταθεί ε, μια διερευνητική επιτροπή. Θα δούμε τι θα αποφασίσει το ILO. Το ζήτημα θα ανακύψει εκ νέου τον επόμενο μήνα και η κυβέρνηση της Γουατεμάλας παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς την κατάσταση για να δούμε ποια μέτρα θα μπορέσουν να ληφθούν. Δεν υπάρχουν εύκολες απαντήσεις. Ναι θα πρέπει να προσαρμοστούμε στις ανάγκες της κάθε χώρας. Ο κύριος Άλλη μίλησε για τις, ε, τη μεγάλη απειλή της τρομοκρατίας στο Πακιστάν. Μιλάμε για πολλαπλούς θανάτους και γι' αυτό η κατάσταση εκεί διαφέρει από τη Βολιβία ή από άλλες χώρες. Βεβαίως αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μικρύνει την εικόνα σε άλλες χώρες. Το θέμα της θανατικής ποινής είναι πολύ σημαντικό. Μιλάμε για 60.000 νεκρούς, αλλά δεν σημαίνει ότι θα ε, βελτιώσουμε την κατάσταση αν σκοτωθούν λίγοι περισσότεροι ή λίγοι λιγότεροι. Αυτή είναι η προσέγγιση πολλές φορές της, Ευρωπαϊκής, ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει να αναγνωρίσουμε τις προκλήσεις και τις διαφορές σε άλλες χώρες. Στη Βολιβία υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα με την εργασία των ανηλίκων. Η Βολιβία λέει ότι εάν το αναγνωρίσουμε τουλάχιστον θα μπορέσουν να έχουν ε, δικαιώματα όπως έχουν όλοι οι εργαζόμενοι. Αν δεν το αναγνωρίσουμε δεν σημαίνει ότι θα απαλληφθεί η παιδική εργασία γιατί η οικογένεια χρειάζεται τα εισοδήματα αυτά αλλά τουλάχιστον να έχουν δικαίωμα στην εκπαίδευση. Αυτό είναι το τέλος του πρώτου γύρου και θα συνεχίσουμε με το δεύτερο Η συνάδελφος αναλαμβάνει την Προεδρία. Thank γνωρίζετε δεν έχουμε πολύ χρόνο, όπως αυτό μας συμβαίνει πάντοτε βέβαια, και αυτό σημαίνει απλώς ότι το θέμα είναι πολύ ενδιαφέρον και ότι υπάρχει μεγάλη ανάγκη συζητήσεως. Τώρα, για να μην απολέσουμε περισσότερο χρόνο, να δώσω τον λόγο αμέσως στο δεύτερο πάνελ, στα πρόσφατα δεύτερο πάνελ. Πρώτα την κυρία Κορίνα Βάργα. Πού βρίσκεστε? Ωραία. Είστε διευθύντρια του Standards Department του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας. Θα εξηγήσετε την άποψη του φορέα monitoring για το GSP. Χρησιμοποιεί η Ευρωπαϊκή Ένωση πλήρω την μόχλευση του GSP συν ή μπορεί να βελτιωθεί. 7 λεπτά. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Εύχομαι καλό απόγευμα σε όλα τα μέλη σας. Ευχαριστώ πρώτα την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου και τον Πρόεδρό της Λάγκε για την ευκαιρία που μας δίνεται σήμερα. Ο ILO χαίρεται για την στρατηγική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που εγκρίθηκε τον προηγούμενο Οκτώβριο που δίνει προτεραιότητα στα διεθνή πρότυπα εργασία στην ατζέντα της για την πρόθεση αξιών. Ο ILO παίζει σημαντικό ρόλο στην πρόθεση των διεθνών αυτών προτύπων και των θεμελιωδών διακυβέρνησης και επίσης βεβαίω υγείας και ασφάλειας των εργαζόμενων δηλαδή. Η εταιρική σχέση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα πλαίσια της εμπορικής της στρατηγικής μπορεί να στηρίξει τις δράσεις του οργανισμού μας και να την καταστήσει, να καταστήσει τις δράσεις αυτές πιο αποτελεσματικές. Ως διευθύντρια του τμήματος προτύπων έχω και άμεση εικόνα του τι σημαίνει για τις χώρες αυτές. Έχω μεγάλη εμπειρία για πολλά χρόνια που έχω εργαστεί επί τόπου, επί του πεδίου δηλαδή, ε, χορηγώντας ε, άμεση εμπειρογνωμοσύνη στις ε, χώρες μέλη. Και τώρα παίζω και τον ενδιάμεσο ρόλο μεταξύ των χωρών και των εποπτικών οργάνων του ILO. Έμαθα πρόσφατα ότι οι προσπάθειε οικοδόμηση δυνατοτήτων μπορούν να εξοικονομήσουν εθνικέ προσπάθειε και εσωτερικώ να ενδυναμώσουν τα εργασιακά πρότυπα στι χώρε δικαιούχου. Ε, εδώ είχα επιπλέον την ευκαιρία να δω ότι αυτά μπορούν να μετατραπούν σε έναν ενάρετο κύκλο με τη βελτίωση των ε, συνθήκων διαβίωσης και με κίνητρα σε εθνικό επίπεδο, αλλά και αντιστρόφως. Δεν χρειάζεται να θυμίσω στην Επιτροπή σας ότι τα διεθνή εργασιακά πρότυπα και τα εποπτικά όργανα του ε, ILO είναι μια βάση για να μπορέσουμε να έχουμε συνολική καθιέρωση των αξιών που μας ενδιαφέρει να επικρατήσουν στον εργασιακό χώρο. Η αξιοπιστία μας είναι γνωστή βάσει των οικονομικών οικουμενικών συμφωνιών για τα εργασιακά πρότυπα και με ένα εύρωστο εποπτικό σύστημα που συνδυάζει ανεξάρτητες ε, και τριμερείς αναλύσεις, ώστε να ακούγεται η φωνή και των επιχειρήσεων και του εργατικού και της κοινωνίας των πολιτών. Ε, το μέρος που ε, επηρεάζεται περισσότερο και ακούγεται λιγότερο κάποιες φορές. Το σύστημα αυτό συνδυάζεται όχι μόνο με την εποπτεία της συμμόρφωσης με τα εργασιακά πρότυπα, αλλά και με την ευθυγράμμιση, με, την, ε, με τις προδιαγραφές τεχνικής συνδρομής του ILO. Αυτά έχουν να κάνουν και με τους οπεπτικούς ε, φορείς και με την κατάσταση κάθε χώρας και προσπαθούμε να βοηθήσουμε στον εντοπισμό των τομέων προτεραιότητας με δράσεις ε, ε, παρακολούθησης και με σενάρια υποθέσεις που να έχουν ωφέλη και προ τι δύο πλευρέ, ώστε να υπάρχει ένα ρυθμό στην επίτευξη των στόχων τη χιλιετία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Οι εποπτικοί φορεί του ILO έχουν συνεισφορέ αναχώρα ε, κατάρτιση συστάσεων και παρακολουθούν την παρακολούθηση των συγκεκριμένων εργασιακών προτύπων στην κάθε χώρα ξεχωριστά για να τονίσουμε τη συνδυασμένη συνολική αυτή προσέγγιση του ILO στην αξιολόγηση, παρακολούθηση και την αποτίμηση, πρέπει εδώ να τονίσω την τεράστια συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πρώτα απ' όλα ως προς τη διαρκή της επαγρύπνηση προκειμένου να παραμένουν προστατευμένα διαρκώς τα εργασιακά δικαιώματα και να συζητούνται και μετά αφιερώνοντας βασικούς πόρους που έχουν ε, βοηθήσει σημαντικά τον ILO να επιτύχει τους στόχους του. Θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας τα ειδικά κίνητρα που έχουν δοθεί για την βιώσιμη ανάπτυξη και την καλή διακυβέρνηση μέσω του συστήματος GSP SYN με μια σειρά από εργαλεία που στις ε, ενδιαφερόμενες χώρες ζητούν να εγκριθούν οι σχετικές συμβάσεις εκ των οποίων οι οκτώ βασικές συμβάσεις του ILO όλο το σύστημα GSP και οι δικαιούχοι του έχουν εκκρεμή ζητήματα που πρέπει να επιληθούν σε σχέση με τις βασικές συμβάσεις του ILO και κάποιες έχουν ε, πολλά κοινά με άλλες χώρες. Ε, εδώ η ειδική αυτή διευθέτηση έχει την ειδική προστιθέμενη αξία να οθεί τις χώρες αυτές προς τη βελτίωση του συστήματο προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αυτό ο στόχο τη διαρκού βελτίωση έχει ανοίξει το δρόμο ώστε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω τη Γενική Διεύθυνση Εμπορίου να στηρίζει την ε, βασική δράση του ΑΕΛΟ σε πολλέ χώρε. Ελσαπαδόρ, Γουατεμάλα, ε, Μογγολία, Πακιστάν. Αυτέ είναι μόνο μερικέ από τι χώρε που τώρα δέχονται τη στήριξή μα με στόχου που θέλουν να αντιμετωπίσουν ζητήματα όπω τη διακριτική μεταχείριση, την καταναγκαστική εργασία, την παιδική εργασία και την ελευθερία του συνασπίζεστε και των συλλογικών διαπραγματεύσεων. Πολλά από τα κοινά μας σχέδια έχουν και την εποπτεία της εργασίας και το ε, επίσημο, την διάσταση της επίσημη εποπτείας, ενώ υπάρχει και οικοδόμηση δυνατοτήτων ώστε να εξασφαλίζουμε την βιωσιμότητα και την συμμετοχή διεθνών εταίρων περαιτέρως, ε, περαιτέρω συμμετοχή θα ζητήσουμε και από άλλες υπηρεσίε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όπως την Γενική Διεύθυνση ΔΕΦΚΟ για να υπάρξει καλύτερη σχέση συνεργασίας μεταξύ ανάπτυξης και ε, εμπορίου και να βελτιωθεί η επιρροή μας, να είναι θετικότερη. Η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων για την σωστή υλοποίηση έχει καλωσορίσει τη μορφή αυτής της συνεργασίας και υπάρχουν συγκεκριμένες απαιτήσει ώστε να συγκεντρωθούν συγκεκριμένες πληροφορίες χώρα που θα πρέπει να μεταφραστούν σε συστάσεις για να αναλυθεί δράση και να περάσουν σε συγκεκριμένα χειροπιαστά μέτρα. Ο ILO θα καλέσει τις δικαιούχους χώρους, χώρες, μεταξύ των οποίων η Αρμενία, ο Παναμάς, η Παραγουάη, οι Φιλιππίνες και το Πράσινο Κροτήρι, να δώσουν ε, μια μεγαλύτερη όθηση στα σχετικά θέματα και βεβαίω με τη στήριξη και την εμπρογνωμοσύνη του ILO. Για να ολοκληρώσω κυρία Πρόεδρε, ο ILO μπορεί μόνο να καλωσορίσει θερμά τι διαδικασίε και τις ε, αποτιμήσεις της Επιτροπής σας σε σχέση με τα θέματα από αξιολόγηση των διεθνών εργασιακών προτύπων με τους ανάλογους οργανισμούς με την ε, συνεισφορά των εποπτικών μηχανισμών ειδικώ με την Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων, την Τριμερή Επιτροπή και την Επιτροπή για τους ε, Συνασπισμούς και Ανώσεις. Εφόσον χρειαστεί μπορεί να, σχηματιστεί και ανακριτική επιτροπή. Σας ευχαριστώ λοιπόν που μου δώσετε αυτή τη δυνατότητα να σας απευθυνθώ και ανυπομονώ για τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ για την ε, προσέλευσή σας και για το γεγονός ότι σεβαστήκατε για το χρόνο αγόρευσή σας. Και τώρα ο λόγος των Στέφαν Βέγγλερ, Πούντος. Α, ωραία. εμπειρογνώμων τελωνιακών θεμάτων για το σύστημα από την Ένωση Εξαγωγικού Εμπορίου. Δεν λειτουργεί το μικρόφωνο του ειδήμονος. Ναι, Πάρ' το πιο κοντά σας, του λέει η κυρία Ρόβολα, αλλά δεν φαίνεται να βοηθεί αυτή η συμβουλή. Sorry, but the microphone doesn't work, even though it... Δεν λειτουργεί το μικρόφωνο, παρόλο που είναι αναμένο το φωτάκι. Να αλλάξετε θέση. Exactly. Perfect. Thank you. So hat das Mikro... Άρα λοιπόν το μικρόφωνο δεν λειτουργούσε από την αρχή. Άρα να αρχίσω από την αρχή τότε. Λέγομαι Βέγγλερ και εκπροσωπώ τα συμφέροντα της εισαγωγικής βιομηχανίας, του εισαγωγικού κλάδου και είμαι και ειδικό για δασμούς στην Foreign Trade Association με έδρα της Βρυξέλλες, η οποία υπάρχει εδώ και 40 χρόνια περίπου και εκπροσωπεί τα συμφέροντα του εισαγωγικού εμπορίου σε ολόκληρη την Ευρώπη, αλλά βεβαίως και παγκοσμίω. Η Foreign Trade Association πιστεύει στο ελεύθερο εμπόριο Free trade, sustainable trade. Δηλαδή βιώσιμο εμπόριο. Γιατί βιώσιμο εμπόριο. Διότι μέσα στα πλαίσια της Free Trade Association επί 12 χρόνια έχουμε την πρωτοβουλία στήριξης πρωτοβουλειών, πρωτοβουλία για την βελτίωση των κοινωνικών προτύπων στις ε, χώρες μέλη. Μπορεί να πει κανείς λοιπόν ότι παλαιότερα που υπήρχε ε, το ελεύθερο παγκόσμιο εμπόριο και τονίζονταν συχνά η αναγκαιότητα του ελεύθερου εμπορίου, αλλά χωρίς βιωσιμότητα ελεύθερο εμπόριο σήμερα στο παγκόσμιο επίπεδο δεν μπορεί να υπάρξει. Στις αρχές της δεκαετίας του 2000 τα πράγματα ήταν διαφορετικά. Όταν δηλαδή τότε επινοήθηκε το σύστημα GSP+, Εκεί τότε το εμπόριο το απέριψε το σύστημα αυτό, διότι θεώρησε ότι δεν συμβαδίζει με τις ανάγκες του εμπορίου και το είχε επικρίνει μάλιστα το σύστημα αυτό, διότι είπαμε τότε ότι μπορεί να οδηγήσει σε στρεβλώσει του ανταγωνισμού. Η άποψη αυτή τα τελευταία χρόνια έχει αλλάξει σημαντικά. Χαιρόμαστε λοιπόν ιδιαίτερα που τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή άρχισε πρωτετραετίας διαβουλεύσεις για ένα νέο σύστημα προτιμήσεων. Έχει εγκύψει το θέμα αυτό, έχει δημιουργήσει ένα σύστημα GSP+, το οποίο πραγματικά αξίζει το όνομα του ως σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων. Γνωρίζουμε επίσης το γεγονό ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά εξ όσων γνωρίζω και οι Ευρωβουλευτές, υποστηρίζουν την εφαρμογή του στις εποφελούμενες χώρες, γιατί με τον τρόπο αυτό όντως βοηθούμε τις χώρες αυτές να βελτιώσουν και την χρηστή διακυβέρνηση και τα δικαιώματα των εργαζόμενων. Έχουμε κατανόηση ότι εφόσον υπάρχουν παραβιάσεις κατά των κανόνων του GSP+, μπορεί η αφαίρεση του καθεστώτος του GSP+, από τη συγκεκριμένη χώρα να είναι ε, ένα ενδεδειγμένο μέτρο. Ωστόσο θεωρούμε ότι πρέπει πριν ε, να φτάσουμε στο μέτρο αυτό να γίνει κάθε δυνατή προσπάθεια για να στηριχτεί η χώρα μέλος, ε, δηλαδή η εποφελούμενη χώρα μέλος, η τρίτη χώρα, να μπορέσει να αποφύγει την ιστατή αυτή ποινή. Διότι οι επιπτώσεις στην ευημερία του πληθυσμού της είναι σημαντικές. Οφείλει κανείς βέβαια να δει ακόμη ότι η προτίμηση των χωρών GPS Plus οδηγεί σε κάποια μειονεκτική μεταχείριση των συνήθων αναπτυσσόμενων χωρών. Οι GSP Plus χώρες και οι χώρες Anything But Arms βρίσκονται και αυτές σε ανταγωνισμό μεταξύ τους. Είναι όμως δύσκολο πραγματικά να εξυπηρετήσει κανείς τα συμφέροντα όλων των χωρών και να θεσπίσει ρυθμίσεις οι οποίες να ανταποκρίνονται ακριβώς στο ενδεχόμενο καθεστώς της κάθε μιας από αυτές τις χώρες. Μπορώ να είμαι σύντομο τώρα σχετικά με τις εμπειρίες του εισαγωγικού εμπορίου. Είναι θετικές. Ποτέ δεν υπήρξε μέχρι τώρα ένα νέο σύστημα, όπως αυτό που θεσπίστηκε προδιετίας, το GSP+, το οποίο να ήταν τόσο θετικά, τόσο καλά διαρθρωμένο και να εφαρμόστηκε τόσο καλά από ε, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και από τις εθνικές τελωνιακές αρχές με τρόπο που πραγματικά να μπορούμε να δηλώσουμε ότι είμαστε απόλυτα ικανοποιημένοι. Και οι εξαγωγικές αναπτυσσόμενες χώρες έδειξαν μεγάλη υπευθυνότητα και φρόντισαν να λειτουργεί το σύστημα GSP Plus χωρίς προσκόμματα. Υπάρχουν βεβαίως κάποιες εξαιρέσεις, αλλά αυτές, ως γνωρίζετε, απλώς επιβεβαιώνουν τον κανόνα. Εν ώψη λοιπόν των θετικών εμπειριών με την εφαρμογή του GSP Plus για την προώθηση της βιωσιμότητας στις αναπτυσσόμενες χώρες, θεωρούμε ότι το GSP Plus θα πρέπει να διατηρηθεί όσο το δυνατόν επί μακρύτερο χρονικό διάστημα. Γιατί δεν εξασφαλίζεται η βιωσιμότητα όταν μια χώρα η οποία βρίσκεται στην φάση των εξετάσεων ας πούμε να μπορεί να διακρίνει ότι πολύ σύντομα μπορεί να χάσει το καθεστώς της χώρας GSP+. Φοβούμε ότι ορισμένες χώρες GSP+, χώρες μέσου εισοδήματος, ενδέχεται, καθώς θα αυξάνει το εισόδημά να εκπέσουν το καθεστώς GSP+. Γρήγορα επιτυγχάνεται το όριο αυτό, ιδίως όταν υπάρχει άνηση κατανομή εισοδήματο μέσα στην χώρα. Για παράδειγμα, η Γκάνα, που δεν είναι χώρα GFP+, έχει αποκλειστεί όμω από το σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων, διότι ο μέσος όρος εισοδήματο είναι πολύ υψηλό. Όμως, το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού τη είναι πάμφτωχο. Λόγω της ανισοκατανομή του εισοδήματο έχασε ωστόσο το καθεστώ τη χώρα μέλους των γενικευμένων προτιμήσεων. Εμείς δεν τα υπέρ της ανύψωσης του επίπεδου. Ζητούμε να ληφθεί η υπόψη η ισοκατανομή του εισοδήματος για να υπάρξει και κάποιο στοιχείο δικαιοσύνης εντός του συστήματος GPS. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ και σας ευχαριστώ, λέει η συμπρόεδρος κ. Ρόβολ, για την τήρηση του χρόνου αγορεύσεως ο κύριος Ρεν Πορτρέν, συντονιστής Justice and Peace. Μάλιστα, σας είδα. Έχει το λόγο αγαπητέ κύριε. Ευχαριστώ πρόεδρε. Η φωνή μου δεν είναι πολύ καλή γιατί ήμουν άρρωστος τις προηγούμενες μέρες Χρειάστηκε να πιω κάτι παραπάνω για να τα καταφέρω. Ε, ζεστά. Ε, είμαι λοιπόν υπεύθυνο ε, για θέματα δικαιοσύνη και ειρήνη στα πλαίσια του συστήματο GSPC. Θα ήθελα εδώ να ε, ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την έκθεση που ετοίμασε. Έχει κάνει τεράστια δουλειά με μια πολύ μικρή ομάδα που στηρίζει και εμένα. Η Ένωση οι ενώσει τη κοινωνία των πολιτών και οι συνδικαλιστικέ οργανώσει παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο για την ε, πρόθεση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, κυρίω των εργασιακών. Και φαίνεται ότι ακριβώ αυτή η φορεί είναι σημαντικότερη για την ε, πρόθεση του συστηματο της GSP-SYN και κάποιες φορές είναι και το πιο δραστήριο μέρος που συμμετέχει στο σύστημα αυτό στις δικαιούχε χώρες. Εμείς ε, από τη δική μας πλευρά, από τη δική μας ε, ένωση, Πιέζουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ασχοληθεί με τα θέματα αυτά και εδώ στις Βρυξέλλες και σε τρίτες χώρες καθ' όλη τη διάρκεια της εφαρμογής του συστήματος GSP. Δηλαδή και κατά την ε, θέσπιση και την υλοποίηση και την παρακολούθηση. Οι απόψεις μας υπάρχουν πολλά διαφορετικά ζητήματα στο πλαίσιο του GSP που θα έπρεπε να διορθωθούν. Τα πρώτα είναι οι ενώσεις της κοινωνίας των πολιτών να συμμετέχουν με τρόπο πιο εύληπτο. Πρέπει να αποσαφινιστεί αυτό. Δεύτερον, Ποιο είναι υπεύθυνο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα θέματα αυτά. Δεν είναι σαφέ για την κοινωνία των πολιτών και τι χώρε δικαιούχου. Για μένα είναι πιο εύκολο γιατί κυκλοφορώ στι Βρυξέλλε, αλλά σε μια δικαιούχο χώρα δεν είναι εύκολο να το καταλάβει κανεί. Τρίτον, Πού συγκεντρώνονται πληροφορίε για τι παραβιάσει και τι βελτιστέ πολιτικέ. Η κοινωνία των πολιτών θέλει να συμμετάσχει, αλλά πού και πώ. Δεν το γνωρίζει. Εδώ λοιπόν θα ήθελα να σταθώ σε τρία ζητήματα. Πρώτα απ' όλα στο θέμα της διαφάνειας, μετά στην ε, συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών και τρίτον στο πώς μπορούμε να βελτιώσουμε την υλοποίηση των συμβάσεων στην πράξη. Θα ξεκινήσω με τη διαφάνεια. Για τις ενώσεις της κοινωνίας των πολιτών παραμένει ασαφές πώς καταμετράται η πρόοδος. Προφανώς έχουμε τις λεγόμενες cards, τα βαθμολόγια που δεν είναι κάτι που διατίθεται στην κοινωνία των πολιτών. Οπότε είτε θα πρέπει να δημοσιοποιούνται αυτά τα βαθμολόγια για να μπορεί να, τα, να λάβει γνώση τους και η κοινωνία των πολιτών, είτε θα πρέπει να συμμετάσχει στην διαδικασία της παρακολούθησης σε αυτό το στάδιο. Ε, παροτρύνουμε λοιπόν εδώ έντονα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δημοσιοποιεί τα βαθμολόγια. Ε, Επίση, δεν είναι σαφέ πόσο πληροφορίε τρίτων μερών μπορεί να διατίθενται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, παρόλο που αυτό ορίζεται από κανονισμό. Η Justice and Peace, λοιπόν, παροτρύνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καθορίσει μια επίσημη διαδικασία αποβολή εκθέσεων για τι ενώσει τη κοινωνία των πολιτών, ώστε να μπορούν να αποβάλουν τι εκθέσει του. Όπω είπε και η κυρία Λοχμπίλερ ήδη, θα μπορούσε αυτό να είναι ένα παράλληλο σύστημα με το σύστημα UPR, που ήδη υπάρχει. Περνάω στο δεύτερο σημείο, η συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών. Παρόλο που το σύστημα GSPC έχει δημιουργηθεί για να βελτιωθούν τα εργασιακά δικαιώματα του εργατικού δυναμικού, οι υπερασπιστές των δικαιωμάτων αυτών ε, από τους φορείς που προανέφερα δεν ε, γίνονται σεβαστές στο δημόσιο χώρο και πολλές φορές ε, γίνονται αντιληπτοί ως απειλές από τις ενδιαφερόμενες κυβερνήσεις. Η συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών, ωστόσο, και των οργανώσεών της χώρες δικαιούχους θα πρέπει να είναι ένας τρόπος για να εξυπηρετηθούν τα συμφέροντα των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων της κοινωνίας των πολιτών και να εξυπηρετηθούν οι κυβερνήσεις στην υλοποίηση των διαφορών συμβάσεων. Θα πρέπει όλοι αυτοί οι φορείς να γίνονται αντιληπτοί ως ένας ισότιμος εταίρος που μπορεί να δημιουργήσει περισσότερες ευκαιρίες στα πλαίσια του συστήματος GSPC. Έτσι, η Justice and Peace παροτρύνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξεύρει μια σφαιρική συνολική προσέγγιση ώστε όλοι οι ε, συμμετέχοντες από την κοινωνία των πολιτών να μπορούν να ασκήσουν πλήρως τα καθήκοντά τους. Αυτό θα μπορούσε να γίνει μέσω της δημιουργίας μιας επιτροπής παρακολούθησης σε μια δικαιούχο χώρα, όπου η κοινωνία των πολιτών θα έχει ένα ρόλο να διαδραματίσει. Επίσης, θα μπορούσε να γίνεται και με εθελούσια συμμετοχή ή σχετικέ συμφωνίε βάσει και του κανονισμού Τίμπερ για την ξυλία. Εδώ θα μπορούσε να υπάρχει και καλύτερη εφαρμογή των συμβάσεων. Αυτό ήταν το τρίτο σημείο που θέλω να αναπτύξω. Η παρακολούθηση είναι πολύ σημαντική για να μην υπάρχει πια ασάφεια όπως προκύπτει τον κανονισμό για το σύστημα GSPC. Θεωρούμε εύστοχο να υπάρξουν συγκεκριμένοι δείκτες ε, συγκριτικής αξιολόγησης, δείκτες οι οποίοι θα είναι χρήσιμοι για να καταμετρήσουμε κάθε πρόοδο ή καθυστέρηση των δικαιούχων χωρών θα μπορούσαμε ακόμη και να σκεφτούμε έναν οδικό χάρτη ε, εφόσον θέλαμε να τον εκπονήσουμε. Επίση, θα μπορούσαν έτσι οι φορεί τη κοινωνία των πολιτών να δραματίσουν ένα ρόλο ε, φύλακα, ε, θεματοφύλακα ε, όλων αυτών των υποχρεώσεων και το κατά πόσο εκπληρώνονται. Οι φορεί τη κοινωνία των πολιτών και η κυβέρνηση που να συνεργάζονται για να προαγκρουθούν τον χώρο των επιχειρήσεων στι δικαιούχε χώρε και να τις υποχρεώνουν να αναλαμβάνουν τι ευθύνε του μετά την υλοποίηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των εργασιακών και των σχετικών συμβάσεων. Ιδίω σε συγκεκριμένου τομεί βλέπουμε ότι αυτό είναι άκρο αναγκαίο. Εν είδη συμπεράσματος. Το εμπόριο με τρίτε χώρε δεν πρέπει να εξυπηρετεί μόνο του πολιτικού και οικονομικού σκοπού τη Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά είναι ένα πολύτιμο εργαλείο για να προωθηθούν τα ανθρώπινα δικαιώματα και δημοκρατία στι χώρε αυτέ. Το σύστημα GSP ΣΥΝ μπορεί να είναι ένα πολύτιμο εργαλείο ώστε να υπάρχει το κατάλληλο πλαίσιο για τις κυβερνήσεις και ε, κατάλληλες διασφαλίσεις για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των εργασιακών. Θα μπορούσε να είναι μια πολύ καλή ευκαιρία εφόσον υπάρχει συνεπή, συνεκτική και σταθερή ε, συμμόρφωση. Γι' αυτό λοιπόν θα επαναλάβω τα βασικά μου σημεία θα έπρεπε να υπάρχει διαφανέστερη πολιτική και υλοποίηση του συστήματος αυτού, να υπάρχει συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών στο όλο πλαίσιο και τέλος να υπάρχουν συγκεκριμένες ε, διαδικασίες κριτικής ε, αξιολόγησης ώστε να καταμετράται σωστά η πρόοδος. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ για την εισήγησή σας και σας ευχαριστούμε που σεβαστήκατε για το χρόνο σας εάν μου επιτρέπετε να πω και κάτι ηρωνικό στην πρότασή σας είναι δύσκολο να γνωρίζουμε ποιος από την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι υπεύθυνο γι' αυτό. Ισχύει για τόσα πολλά πράγματα. Σας ευχαριστώ πολύ που το επαναλάβατε. Δεν ισχύει μόνο για τον GSPC αυτό. Ο λόγος στον Ζαχούρ Αγουάν, πρόεδρο της ε, Σύνομοσπονδίας Εργαζομένων του Πακιστάν. Ε, υπάρχουν πολλοί λόγοι για να σας δώσει κανείς το λόγο, αλλά πρωτίστως σας τον δίνουμε, διότι θεωρούμε ότι είναι σημαντικό να ακούσουμε κάποιον εκπρόσωπο της κοινωνίας των πολιτών από μια τέτοια χώρα. Χώρα που έχει ολοκληρώσει τη διαδικασία αξιολόγησης, χώρα που έχει καταβάλει έντονες προσπάθειες για να συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις όπως προκύπτουν από τις διεθνείς συμβάσεις. Σε πολλά μέρη του κόσμου η κοινωνία των πολιτών δεν έχει την ελευθερία να εκφραστεί όπως θα ήθελε, οπότε παρακαλούμε εκφραστείτε εδώ. Σας δίνω το λόγο που είστε. Α, ωραία. Ε, thanks, Madam Chair. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ επίσης και την Επιτροπή γιατί κάλεσε τη Συνομοσπονδία Εργατών, ένα σημαντικό πυλώνα της κοινωνίας των πολιτών και είμαι ευγνώμων προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και το γραφείο της Κομισιόν στο Πακιστάν γιατί βρίσκεται σε συνεχή επαφή μαζί μας για να δούμε πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τις συνθήκες εργασίας και διαβίωσης στο Πακιστάν, διότι από τις 27 συμβάσεις των γενικευμένων προτιμήσεων, 16 αφορούν το εργατικό δυναμικό καθώς και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Μιλάμε για 60 εκατομμύρια εργατικό δυναμικό. Και καταλαβαίνετε ότι και αν λάβουμε υπόψη και τα άλλα μέλη του νοικοκυριού, τότε συμμετέχουν στο εργατικό δυναμικό, συμμετέχει το 90% του πληθυσμού. Ελπίζω λοιπόν να μπορέσετε να μας ε, δώσετε ένα feedback που ε, χρειαζόμαστε, κάτι το οποίο προανέφερε και ο κύριος Άλλη. Και αυτό που μας βοήθησε ήταν ότι συμμετείχαν όλες τις περιφέρειες του Πακιστάν και οι υπεύθυνοι για ζητήματα εργατικού δυναμικού και στο Υπουργικό Συμβούλιο. Συμφωνούμε με την Επιτροπή γιατί τονίσαμε πτυχές που, στις οποίες έχει αναφερθεί και η Κομισιόν. Ποια είναι δηλαδή τα, τα προβλήματα του εργατικού δυναμικού στη χώρα μας. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι τι απομένει να εφαρμοστεί για τα επόμενα χρόνια, γιατί μιλάμε για ένα διετές ε, πλαίσιο μέχρι ε, τώρα. Θα ήθελα να αναφερθώ στους τέσσερους, στους τέσσερις ε, τομείς βασικούς τιμής, τομείς δηλαδή ε, στην εργασία των ανηλίκων, στο εργατικό δυναμικό και στις ε, συλλογικές διαπραγματεύσεις καθώς και την εργασία των ανηλίκων. Μιλούσαμε για 3,3 εκατομμύρια εργασία ανηλίκων. Αυτό δείχνει η μελέτη, αλλά τώρα μιλάμε για 2,7 εκατομμύρια και μειώνεται ο αριθμός της εργασίας ανηλίκων, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι υπάρχει ένα ε, θέμα δημογραφικής ανάπτυξης πάρα πολύ γρήγορης μετά από την Ινδία και την Αυστραλία. Άρα καταβάλλεται προσπάθεια να αντιμετωπίσουμε αυτό το ζήτημα και να εφαρμόσουμε τα σωστά δεδομένα. Και το Παντζάμπ έχει κάνει ρηξικέλευτα βήματα, ιδιαίτερα στον τομέα της εκπαίδευσης, που αποτελεί το ίμιση της επικράτειας του Πακιστάν σε σχέση με το εργατικό δυναμικό και το επίπεδο του εργατικού, δυναμικού, αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να δούμε τι γίνεται στις ε, βιομηχανίες και ιδιαίτερα όταν οι εργαζόμενοι δεν έχουν τη σωστή ασφάλεια. Θα πρέπει να υπάρχουν σωστές κοινωνικές προδιαγραφές και δίχτυα ασφαλείας, διότι πολλές φορές ε, δυστυχώς οι εργαζόμενοι δεν εντάσσονται σε ένα ασφαλιστικό σχήμα. Μόνο δίκο το 20% εντάσσεται σε αυτό το πλαίσιο ασφάλισης. Έχουν γίνει βεβαίως ε, πρόοδοι, αλλά δεν θα ήθελα να μπω σε λεπτομέρειες. Ως προς τις διακρίσεις, λέμε ότι οι δύο ε, περιφέρειες, το Πάντζαπ και μία άλλη, έχουν ενταχθεί σε αυτό το πλαίσιο και δεν ακολουθούν ταχεία βήματα. Υπάρχει λοιπόν δυστυχώς διάκριση σε επίπεδο της αγοράς εργασίας και νομίζω ότι υπάρχουν διαφορετικά νομοθετικά πλαίσια από τις περιφέρειες πέρα από το ε, θέμα της ε, εργασίας ανηλίκων. Ως προς τις συλλογικές συμβάσεις και τις συλλογικές διαπραγματεύσεις θα πρέπει να λειτουργήσουν σωστά τα συνδικάτα για να μπορούμε να φτάσουμε σε συλλογικές διαπραγματεύσεις και συμφωνήσεις, συμφωνίες, με συγχωρείτε. Και αυτό που έχει σημασία είναι να μην υπάρχουν διακρίσεις φύλων, να μην υπάρχει εργασία ανηλίκων και να υπάρχουν και συλλογικές διαπραγματεύσεις και συμφωνίες. Θα πρέπει να δούμε ότι στον ιδιωτικό τομέα είναι πολύ δύσκολο να δράσουν τα συνδικάτα και υπάρχουν ε, συνδικάτα σε ένα επίπεδο 4% ε, σε εθνικό επίπεδο. Σε επίπεδο αγροτικής οικονομίας δεν υπάρχει καθόλου συνδικαλισμός. Και αυτό που έχει σημασία είναι να υπάρχει και επιθεώρηση εργασίας που δεν υπάρχει. Και αυτό που έχει σημασία είναι ότι για 351.000 επιχειρήσεις υπάρχουν μόνο 427 επιθεωρητές. Άρα δεν υπάρχει ένα σωστό ε, δείγμα ασφάλειας. Υπάρχει μία έκθεση πρόοδου την οποία σας δείχνω έτσι ώστε να υπάρχει σωστότερη συμμόρφωση. Αλλά επειδή δεν έχω χρόνο δεν θα επεκταθώ. Θα ήθελα να πω ότι όχι μόνο στο Πακιστάν αλλά και σε άλλες χώρες υπάρχει μεγάλο πρόβλημα ως προς την εφαρμογή των νόμων μέσα στα πλαίσια των ε, γενικευμένων προτιμήσεων και των ευεργετούμενων χωρών. Αυτό που μας ε, ενδιαφέρει είναι να δούμε κατά πόσο υπάρχει εκμετάλλευση των εργαζομένων. Υπάρχουν πολλαπλά κέρδη για πολύ λίγους. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι, μεγάλοι, οι μεγάλες επιχειρήσεις δεν επιτρέπουν στους εργαζόμενους να μπορέσουν να ζήσουν καλά τη ζωή τους και να μπορέσουν να συμμετάσχουν σωστά στο, παραγωγικό, στην παραγωγική αλυσίδα. Γι' αυτό υπάρχουν μεγάλες θυσίες ως προς τα ανθρώπινα δικαιώματα το συνδικαλίζεστε, το δικαίωμα του συνδικαλίζεστε και το δικαίωμα των συλλογικών διαπραγματεύσεων, τα οποία παραβιάζονται. Θα πρέπει λοιπόν να καταβάλουμε κάθε προσπάθεια να βελτιώσουμε και τους τρεις αυτούς τομείς. Thank Έχουμε λοιπόν χρόνο για μια σειρά ερωτήσεων. Και μετά θα δώσω το λόγο πάλι στους πάνελιστ για να απαντήσουν ενδεχομένως και να σχολιάσουν. Έχουμε 32 λεπτά έως και 31 στη διάθεσή μας. Ε, ο εισηγητής δεν είναι εδώ. Η Σκά Κέλλερ έχει το λόγο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους ομιλητές. Σας ευχαριστούμε που ήρθατε και μας είπατε τις απόψεις σας. Έχω μια-δυο ερωτήσεις προς τους διάφορους παρεμβαίνοντες. Προς τον εκπρόσωπο του ΕΛΟ θέλω να ρωτήσω εάν θεωρείτε ότι μπορεί να βελτιωθεί από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης η όλη υλοποίηση των συστάσεων του ΕΛΟ. Βεβαίω αναφέρονται διαρκώ σχετικέ εκθέσει, όμω θεωρείτε ότι μπορούσαμε να κάνουμε περισσότερο ω έκθεση, ω ε, Ευρωπαϊκή Ένωση. Κατά τα άλλα, νομίζω από το ε, Justice and Peace ε, έχετε ξανακάνει ανάλογε προτάσει. Τα είπαμε χθε και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν είναι εδώ η εκπροσωπή τη. Και τώρα η ερώτησή μου ουσιαστικά στρέφεται προ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πώ τη συζητάμε αυτέ τι προτάσει, Μιλάμε για προτάσεις που σας κάνουν οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις. Τις έχετε ακούσει, τις έχετε καταγράψει, έχετε ήδη αρχίσει να τις εφαρμόζετε, πώς. Έπειτα προς τον κύριο Εουάν, ευχαριστούμε που ήρθατε και πολύ πρακτικά. Μιας και μιλάμε για κοινωνικό διάλογο και ενδιαφερομένους συμμετέχοντες κτλ. Πόσο Πολλοί συμμετέχετε στο Πακιστάν στα πράγματα αυτά. Συμμετέχετε με την πρόσκληση και άλλων φορέων της κοινωνίας των πολιτών. Λαμβάνετε υπόψη δική σας προοπτική, οι απόψη σας, οι προτάσεις σας. Έχετε συνολικά την αίσθηση ότι η δική σας η προοπτική γίνεται σεβαστή. Θα περιμένατε περισσότερα. Πώς είναι στην πράξη η συνεργασία σας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό θα μας ενδιέφερε. Και επίσης και αυτό είναι κάπως ευρύτερο, τι άποψη έχετε για τη συνεργασία σας με τους εργοδότες, το όλο σύστημα GSP Plus, πώς μπορεί να προστατεύσει τα δικαιώματα εργαζομένων και εργοδοτών ταυτόχρονα. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Μόσχα. Ευχαριστώ. Μια γενική ερώτηση προς όλους τους παρεμβαίνοντες. Διότι όταν συμμετέχουμε σε τέτοιου είδους ακροάσεις, Τελικώς, αυτό που γίνεται σαφές στο τέλος είναι ότι η μετάβαση από την παρακολούθηση στην υλοποίηση και στην επίτευξη συγκεκριμένης πρόοδου χειροπιαστής είναι το αδύναμο σημείο, το στάδιο αυτό που ακριβώς δεν υπάρχει ένα συγκεκριμένο μοντέλο και που θα έπρεπε ίσως να προσαρμοστεί τις ανάγκες κάθε χώρας ανάλογα με τις φορές που επικρατούν. Όμως θα έπρεπε να υπάρχει και μια συλλογή βελτιστών πρακτικών όπως ακούστηκε για να διευκολυνθούν και όσοι στην πράξη κάνουν την πρακτική δουλειά. Μία συγκεκριμένη συνεισφορά στο πώς να προσαρμοστούν οι πράξεις που πρέπει να υλοποιηθούν. Ερωτώ λοιπόν τους ομιλητές μας, τι είδους παρέμβαση ήταν χρήσιμη, τι είδους συλλογή πληροφοριών, πώς θα μπορούσαν αυτά να πάρουν σάρκα και οστά σε πραγματικές βέλτιστες πρακτικές και πώς θα μπορούσαμε κι εμείς να διευκολυνθούμε ώστε να αξιοποιούμε καλύτερα και να έχουμε μέτρα τα οποία είναι πιο συγκεκριμένα και ξεπερνούν απλώς την έκφραση απόψεων για τις νομοθετικές τροποποίησεις. Γιατί όπως ξέρουμε νομοθετικές τροποποίησεις είναι κάτι που μπορεί κανείς να το δει, να το καταμετρήσει, αλλά είναι απλώς ένα από τα πρωταρχικότερα στάδια όλες τις δουλειά που πρέπει να γίνει. Διερωτώμε λοιπόν, μπορεί να δημιουργηθεί ένα μοντέλο για τα εργαλεία συγκεκριμένη αξιολόγηση και αυτά μπορούν να μεταφραστούν σε δουλειά της Επιτροπής που θα το πάρει το μοντέλο αυτό και θα το κάνει πράξη στις διάφορες χώρες, μία-μία. Ευχαριστούμε πολύ. Α, κύριε Ντάρλινγκ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Έχω μια παρόμοια ερώτηση όπως αυτή της κυρίας Μόσκα σχετικά με το τι μπορεί να γίνει για τη βελτίωση. Όμως έχω και μια ιδιαίτερη ερώτηση για τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου. Και μετά τα όσα είπε ο κ. Άουαν, πολύ ε, εντυπωσιακά αυτά. Ποια είναι η δική σας εντύπωση σε ό,τι αφορά την εφαρμογή των προτύπων στις εξαγωγές αφού γνωρίζουμε ότι οι εξαγωγέ χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο από αναπτυσσόμενε χώρε σε σχέση με την Ευρώπη. Χρειαζόμαστε ειδικά προγράμματα σε ό,τι αφορά τι ε, εξαγωγικέ ζώνε. Τα δικαιώματα των εργαζόμενων γίνονται σεβαστά στην, ε, στις εξαγωγικές ζώνες. Ε, από την εμπειρία μου ως συνδικαλίστρια ηγέτης έχω ακούσει φρικτά πράγματα για αυτά. Είναι δυνατόν λοιπόν να βελτιώσουμε την κατάσταση διαβίωσης μεγάλων μέρων, μεγάλου μέρους του πληθυσμού. Η υποβάθμιση εργατικών δικαιωμάτων εφόσον συμβαδίζει με αυτήν την προσπάθεια βελτίωσης δηλαδή σε ορισμένες περιοχές και ιδίω αναφέρομαι βέβαια στην ε, αρχή της ελευθερίας του συνεταιρίζεστε και ε, τις συνδικαλιστικές ελευθερίες. Ο Μπεν Ευχαριστώ. Πρώτα. Ερώτηση για τον κύριο Βέγγλερ. Γίνεται όλο και πιο ενδιαφέρον συζήτηση αυτών των supply chains, των αλυσίδων προμηθειών είναι αποδεκτές εκεί οι συνθήκες, ιδίως για τα υφαντουργικά προϊόντα. Εκεί η συμμετοχή της συγκεκριμένη χώρας στην GSP SIN παίζει κάποιο ρόλο για τις επιχειρήσεις που εξάγουν ώστε δηλαδή να μπορούν να τα αποκρίνονται και περισσότερο στις προσδοκίες των καταναλωτών. Και μία ερώτηση με τον κύριο Άουαν αυτή η ανεξάρτητη έκθεση για το GSP Plus μου φαίνεται πραγματικά σημαντική και νομίζω ότι είναι και μοναδική παγκοσμίω. Ποιες ήταν οι προκλήσεις για την σύνταξη εκθέσεως αυτής. Μπορείτε να το εξηγήσετε. Βεβαίως αυτά τα πράγματα κοστίζουν και χρήματα. Μήπως μπορούμε έτσι δηλαδή να σπρώξουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να χορηγήσει κίνητρα και προς άλλους, σε άλλες χώρες να κάνουν κάτι παρόμοιο η πρόεδρος Ρόβολ. Άλλοι οι οποίοι επιθυμούν να συζητήσουν ή να θέσουν ερωτήσεις. Αμέσως, αμέσως θα σας δώσω το λόγο. Έχω μια ερώτηση προς όλες και όλους τους συμμετέχοντες. Πώς μπορεί να διασφαλιστεί ώστε τα συμφωνημένα να φτάσουν πραγματικά να ωφελήσουν τους εργαζόμενους στις επιχειρήσεις επιτόπου. Έχω κάπως κάποιες αμφιβολίες ότι ωραία τα λέμε εδώ, ωραίες αποφάσεις λαμβάνουμε, αλλά στο τέλος της αλυσίδας τα πράγματα ίσως δίνουν μια διαφορετική εικόνα. Αυτή ήταν μια ερώτηση γενικού χαρακτήρως. Θα έλεγα τώρα ότι υπάρχει εκπρόσωπος θήλεως γένους της Ινδονησίας. Είστε εσείς κυρία μου. Ωραία. Και μετά θα δώσω πάλι το λόγο στα μέλη του πάνελ. Ε, ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, λέγομαι Σεγκάφτ και είμαι βουλευτής από το Ινδονησιακό Κοινοβούλιο. Είναι μεγάλη τιμή για μένα και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω κιόλας για την πρόσκλησή σας. Βρισκόμαστε εδώ για τις συναντήσεις του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου. Μάθαμε πολλά από την έκθεσή σας και εκτιμούμε πολύ το περιεχόμενό της. Θα ήθελα μάλιστα να θέσω μια ερώτηση προς εσάς, δηλαδή τα μέλη της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου. Η Ινδονησία υποδέχεται, υποδέχεται την επόμενη συνάντηση των Υπουργών Εμπορίου του ΠΟΕ και παραλλήλως θα συνεδριάσουν και εκπρόσωποι Τη κοινωνία των πολιτών. Έχουμε το, τη δέση μέτρων του Μπάλι για το λεγόμενο Public Stock Holding. Και στο 2015 στο Ναϊρόμπι οι υπουργοί συμφώνησαν να το εφαρμόσουν μέχρι το 2017. Η δική μου λοιπόν ερώτηση έχει ως εξής. Πώς συνδυάζεται το έργο σας στην Κοινοβουλευτική σας Επιτροπή για την εφαρμογή του θέματος αυτού για τη βελτίωση της ευημερίας των ανθρώπων. Εμείς, η Ινδονησιακή λοιπόν Εθνοσυνέλευση, έχει, έχουμε φτιάξει μια ειδική task force που εγκύπτει σε θέματα στόχων της χιλιετίας έτσι ώστε να μην ξεστρατήσουν εντός εισαγωγικών οι προσπάθειες για την εφαρμογή των στόχων αυτών. Ευχαριστώ. Τώρα λοιπόν θα προχωρήσουμε με αντίστροφη σειρά. Πρώτα θα ακούσουμε τον κύριο Άουαν. Μπορείτε να σχολιάσετε. Ε, Ευχαριστώ Πρόεδρε. Για να πω την αλήθεια, η πρώτη ε, ερώτηση έχει να κάνει με τον κοινωνικό διάλογο σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ενώσης και πώς μπορεί αυτό να γίνει και στο Ισλαμαπάντ με τον εκπρόσωπο τον είπα όταν πρώτα απ' όλα ξανασυζητιέται το σύστημα GSPC ε, προσκλήθηκαν οι συνδικαλιστικές οργανώσεις για να το συζητήσουμε αυτό και ακούστηκε η φορά των εργαζομένων. Όμως, ε, παρόλο που είμαστε ευγνώμονες που υπήρξε πριν τη δημοσιοποίηση της έκθεσης διαβούλευση με τους συνδικαλιστές, έγιναν κάποιες συναντήσεις και Μας βοήθησαν και οι ανάλογες ενώσεις εδώ στις Βρυξέλλες, ε, κυρίως της γερμανικής σύνθεσης. Όμως ο κοινωνικός διαλόγος χρειάζεται για να έχουμε και τους κατάλληλους μηχανισμούς. Ίσως οι άνθρωποι της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και οι ίδιοι γνωρίζουν πολύ καλά ότι θα έπρεπε να υπάρχει κοινωνικό διάλογο. Όμω, νομίζω ότι όσο και αν είμαστε ευγνώμονε, δεν ήταν τελικά υπαρκτό ο μηχανισμό. Υπάρχει όμω ανάγκη για τέτοιο μηχανισμό. Χρειάζεται γιατί ε, όπου έχει γραφεί η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να υπάρχει ο ανάλογος συσχετισμός και κυρίως σε συνδυασμό με τις ενώσεις των, των εργαζομένων. Υπάρχουν συγκεκριμένε συνδρομές, ευθύνες στα πλαίσια του ILO, υπάρχει αιτήσια καταμέτρηση της προόδου, της συμμετοχής των συνδικαλιστικών οργανώσεων. Τα είναι τα κομβικά σημεία για να γίνει βελτίωση στις εργασιακές συνθήκες και της συνθήκες διαβίωσης. Οι σχέσεις με τους εργοδότες. Έχουμε πολύ καλό κοινωνικό διάλογο και είμαστε μια από τις μόνες χώρες που έχουμε την πρωτιά να έχουμε με τους πεφωτισμένους εργοδότες ένα συμβούλιο δίμερες με συμμετοχή και εργαζομένων και εργοδοτών όπου φύγονται όλα αυτά τα θέματα. Τη στιγμή που ξεκινούσε η πόνηση τη έκθεση αυτή, ήταν και η κυρία Νταλή και ο υπεύθυνο για τα περιφερειακά θέματα του Πακιστάν, ε, τότε ναι, εντοπίσαμε προβλήματα με κάποιους εργοδότες που δεν είχαν ε, καταγραφεί, δεν ήταν νόμιμοι. Και το πρόβλημά του ήταν πόσο περισσότερη εξουσία θα μπορούσαν να πάρουν. Την άρπαζαν όποτε μπορούσαν η εφαρμογή του εργατικού δικαίου ήταν θέμα αυθαίρετο κάθε επιχείρηση. Οπότε ο κάθε εργαζόμενο κοίταζε όχι πώ εφαρμόζεται το εργατικό δίκαιο, αλλά αν έπαιρνε ένα αξιοπρεπή μισθό σε πρώτη φάση. Δεν υπήρχε λοιπόν ακριβώ η σωστή διαδικασία. Σε κάποιε περιπτώσει δεν υπήρχαν όμω καν συνδικαλιστικέ οργανώσει για να εκπροσωπήσουν του εργαζομένου. Για τα προβλήματα λοιπόν, όπως καταγράφονται στην έκθεση, παρόλο που νομίζω ότι μεγάλο μέρος της έκθεσης ε, εκπονήθηκε από εμά τους ίδιους, αλλά μόνο και μόνο για την μελέτη, είχαμε α, την συμμετοχή της γερμανικής ε, ε, ομολόγου μας Ένωσης. Γι' αυτό μπορέσαμε να τα καταρτήσουμε αυτά. Χρειάζεται πάντως περισσότερη παρακολούθηση, περισσότερη ευαισθητοποίηση στο Πακιστάν σε θέματα όπως αυτή η έκθεση. Χαίρομαι πάντως που μπορούσατε να τα έχετε. Είναι ε, κάτι που μπορεί να κάνει κάθε συνδικαλιστική οργάνωση. Ελευθερώνονται περισσότερες προσπάθειες από τους ενδιαφερομένους και τους συμμετέχοντες. Όταν λέμε βιώσιμη ανάπτυξη, πώς να τη βιώσουμε αυτή τη βιώσιμη ανάπτυξη. Όταν λέμε GSP απαιτεί οικοδόμηση δυνατοτήτων για όλους τους ε, ενδιαφερομένους ε, και για τους ε, συνδικαλιστές βεβαίως, αλλά και για τις κυβερνήσεις. Και αυτοί πρέπει να κάνουν κάτι. Από την πλευρά λοιπόν των εργαζομένων, ε, βεβαίω το θέμα τη εργασία το έχουν αναλάβει περιφέρειες. Πρέπει να δούμε ποιε είναι καθυστερημένε στο Πακιστάν, ποιε είναι πιο μπροστά και πρέπει κυρίω να υπάρξει οικοδόμηση δυνατοτήτων για τις ε, περιφερειές αυτές, για να προχωρήσουν και αυτές. Και πρέπει να υπάρχει οικοδόμηση δυνατοτήτων ε, πρέπει να υπάρξει λοιπόν προσπάθεια προόδου και από τις κυβερνήσεις για να υπάρξει μια αρμονική συνολική εικόνα. Και τέλος, όταν είπατε για αυτές τις supply chains και τα λοιπά, αυτοί οι πολυεθνικοί παγκόσμιοι κανόνες πόσα παίρνει ο διάμεσος, πόσα προσπαθεί να κάνει, τι γίνεται στο τέλος. Υπάρχει πολύ μεγαλύτερη διαφορά στην ουσία και πρέπει να καταλάβουμε ότι βρισκόμαστε στον 21ο αιώνα. Στον 21ο αιώνα παρά τα θεαματικά ε, πρώτη θεαματική άνοδο του παγκόσμιου εισοδήματο, ένα πέμπτο του παγκόσμιου πληθυσμού ε, πηγαίνει να κοιμηθεί πεινασμένο και ζουν σε άθλιες συνθήκες ε, σε συνθήκες όπως αυτές που ίσχυαν παντού πριν από 100 ε, χρόνια στην πόλη του Σικάγο που τους ανάγκασαν να βγουν στους δρόμους, να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους αλλά που οδήγησαν και σε θυσίες που έφεραν καλύτερες ζωές. Σας ευχαριστώ να σταθώ στο θέμα της υλοποίησης που νομίζω ότι ήταν η ερώτηση που τέθηκε από όλους. Δεδομένης της ποικιλία της νομοθεσία μεταξύ των δικαιούχων χωρών δεν υπάρχει ένα συγκεκριμένο αποτύπωμα που θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει ο καθένας για όλους. Η κάθε μια έχει τις ιδιαιτερότητές της. Όμως υπάρχουν τοπικές επιτροπές της κοινωνίας των πολιτών, των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, των επιχειρήσεων, των κυβερνήσεων που θα μπορούσαν να μας επιτρέψουν να δημιουργήσουμε ένα ε, σχέδιο δράσης για το πώς να προωθήσουμε την υλοποίηση των συμβάσεων. Αυτά απαιτούν και την χρήση δικτών συγκριτικής αξιολόγησης. Benchmarks οι οποίοι να βασίζονται στο κατά πόσο είναι εφικτοί. Εάν δεν συμμετέχουν όλοι γύρω από ένα τραπέζι συζήτησης δεν θα προχωρήσει το πράγμα. Επιπλέον, ε, για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία και το πρόγραμμα δράση ε, του ΟΗΕ ε, δηλώνεται και αυτό. Πρέπει να, να διευκολυνθεί ο κοινωνικό διάλογο. Πρέπει αυτό το πολιτικό εργαλείο να το χρησιμοποιήσουμε για να πιέσουμε υπέρ του κοινωνικού διαλόγου στι χώρε δικαιούχου των GSP. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Επόμενο. Στέφαν Βέγγλερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Απαντώ σύντομα στο ερώτημα του κυρίου Λάνγκε. Εάν οι χώρες του GPS Plus προσφέρουν και κίνητρο να αγοράζει κανείς προϊόντα τους. Η απάντηση είναι σαφώς καταφατική. Επιχειρήσεις οι οποίες μετακινούν την παραγωγή τους σε τέτοιες χώρες, εφόσον υπάρχει ο κίνδυνος να αφαιρεθεί πάλι το καθεστώς ε, το GSP Plus, μπορεί να είναι πολύ υψηλός. ασφαλώς εποφελείται και ο καταναλωτής. Όποιες επιχειρήσεις δεν αγοράζουν από τις χώρες αυτές λόγω των υψηλών προτύπων, ας μην λησμονούν ότι οι χώρες αυτές έχουν υπογράψει το εάν τηρούνται τα πράγματα αυτά από τις επιχειρήσεις είναι άλλη υπόθεση. Και με το σύστημα Business Social Compliance έχουμε συλλέξει την εμπειρία ότι πρέπει να ενισχυθεί η συνείδηση, η ευαισθητοποίηση υπέρ των κοινωνικών προτύπων. Διότι αν αρχίσουν καλά και μετά από κάποια χρόνια ξαναρχίσουν οι ατασταλίες, τότε το πράγμα δεν προχωρεί καλά. Ευχαριστώ και ευχαριστώ για τις ερωτήσεις σας. Για την πρώτη ερώτηση, αν η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να πράξει περισσότερα για να προωθήσει τις συνθήκες του ILO. Και μόνο το γεγονός ότι δίνονται, δίνεται προτεραιότητα στο θεματολόγιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μια εμπορική πολιτική βασισμένη σε αξίες έχει παίξει σημαντικό ρόλο. Η συνεργασία μας στον τομέα αυτό είναι σχετικά νέα. Αρχίσαμε με λίγες χώρες και επεκτηνόμαστε σε περισσότερες. Υπάρχει λοιπόν χώρος για επέκταση της συνεργασίας Ιδίω σε επίπεδο χωρών. Ήδη ενημερώνουμε και εκπαιδεύουμε τους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις διάφορες χώρες για το πώς λειτουργεί το σύστημα. Αυτό έχει σημασία για τους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις χώρες αυτές για να κατανοήσουν καλύτερα πώς λειτουργούν τα συστήματα κοινωνικά και άλλα εκεί και ασφαλώς θα συνεχίσουμε να το πράττουμε για να διασφαλίσουμε ώστε οι αντιπροσωπείες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο επίπεδο των χωρών εταίρων να μπορούν να είναι και συνομιλητής μας στο αναγκαίο επίπεδο. Αν μπορούν να γίνουν και άλλα πράγματα, βεβαίως πάντα μπορούν να γίνουν και άλλα πράγματα. Μπορούμε να επεκτείνουμε λοιπόν συνεργασία από την άποψη αυτή. Δεύτερο, ο αδύναμος κρίκος που είναι η εφαρμογή. Όντως, ναι, από εκεί προκύπτουν οι περισσότερες προκλήσεις όταν ξεφεύγουμε πλέον από τα θεωρητικά κείμενα και μπαίνουμε στην πραγματική ζωή. Εδώ ωστόσο για τις βέλτιστες πρακτικές και μιλώ για την διάσταση των εργατικών δικαιωμάτων έχουμε καλή απήχηση ιδίως σε θέματα παιδικής εργασίας όπου έχει καταβάλει σημαντικές προσπάθειες ο ΑΕΛΟ τα τελευταία 20 χρόνια. Ξέρουμε λοιπόν ποια πράγματα λειτουργούν καλά, ξέρουμε πώς να επιτύχουμε περισσότερη απήχηση. Βεβαίως, τα νούμερα είναι ακόμα επιβαρυντικά για το Πακιστάν, όμως κινούνται προς την κατεύθυνση. Έχουμε και κάποιες ορθές πρακτικές σε κάποιους τομείς. Κάτι που αξίζει να του χαρίσετε περισσότερη προσοχή είναι ο χώρος των διακρίσεων, όπου εκεί μας λείπουν και βασικά δεδομένα και βεβαίως και ορθές πρακτικές. Και ο δεύτερο τομέας που θέλω να τονίσω και όπου όπου όλοι μπορούμε να επιφέρουμε μια βελτίωση είναι οι επιπτώσεις των πολιτικών αυτών. Εκεί όπου μπορούμε επίσης να κάνουμε προσπάθεια, όπου δηλαδή αποκλείονται κάποιοι από την εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας, εκεί υπάρχει ένα σημαντικό πρόβλημα, το ίδιο και η πρόσβαση επιθεωρητών, που καμιά φορά παρεμποδίζονται. Ο εποπτικός φορέας του ILO έχει δώσει ιδιαίτερη σημασία σε αυτά. Επίσης να φροντίσουμε ώστε όλα όσα συμφωνούμε να εφαρμόζονται στις συγκεκριμένες χώρες. Το τονίζω και εγώ αυτό. Τέλος, το εποπτικό σύστημα του ILO αυτό παρακολουθεί σε τακτική βάση. Ότι τα όσα συμφωνούνται και κυρώνονται σε ό,τι αφορά τα εργατικά δικαιώματα να εφαρμόζονται και πράγματι στην πράξη. Και ένα άλλο σημαντικό γεγονός που επιθυμώ να τονίσω είναι να έχουν και οι συνδικαλιστές της επιχειρήσης πρόσβαση στο εποπτικό σύστημα, να μπορούν να υποβάλουν δηλαδή αναφορές, εκθέσεις και με τον τρόπο αυτό να έχει και η κοινωνία των πολιτών πρόσβαση στο εποπτικό σύστημα. Το εποπτικό σύστημα το ΙΕΛΟ να μην βασίζεται μονάχα σε εκθέσεις που λαμβάνει από τις κυβερνήσεις, αλλά και σε αναφορές κάθετα εκθέσεις, που λαμβάνει και από φορείς της κοινωνίας των πολιτών. Αυτά σας ευχαριστώ. Ας λάβει το λόγο τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να προβεί σε αξιολόγηση, να μπορέσει να απαντήσει και σε άλλες ερωτήσεις αν είναι δυνατόν. Εξ όσων βλέπω εδώ έχουμε κοντά μας την Διευθύντρια της Digitrade Σάντρα Καλίνα. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα καταρχήν να σας ευχαριστήσω για αυτό το ιδιαίτερα, ε, το εξαιρετικό απόγευμα, γιατί μας δώσατε τροφή για σκέψη. Όταν αρχίσαμε να εφαρμόσουμε το GSP, τις γενικευμένες προτιμήσεις ε, πρόπερση δεν είχαμε οδηγίες χρήσης. Δεν ξέραμε πώς να αρχίσουμε αυτή την επεξεργασία. Γι' αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω τον πρόεδρο Λάγκε γιατί άρχισε, αρχίσαμε μαζί με το ILO να ε, ορίσουμε αυτό το ενιολογικό σύστημα. Δηλαδή αρχίσαμε αυτό το εγχείρημα χωρίς να ξέρουμε πώς θα το χειριστούμε έμπρακτα. Ως προς τη διαφάνεια ξέρετε ότι μας ενδιαφέρει άμεσα, γι' αυτό και ε, για πρώτη φορά ερμηνεύεται και εκδίδεται αυτή η έκθεση την οποία θα μετρήσουμε σε σχέση με την επόμενη. Και έτσι θα μπορέσουμε να οριοθετήσουμε το όλο πλαίσιο και να έχουμε ορόσημα. Θα ήθελα να πω ότι χαίρομαι γιατί υπάρχει σαφής ε, διάλογος με την κοινωνία των πολιτών. Μιλήσαμε και με τον εκπρόσωπο του Justice and Peace. Αυτό όμως ε, δεν είναι καθόλου μικρό υπεριορισμένο ε, κατόρθωμα. Ακούσαμε και από το Διεθνή Οργανισμό Εργασίας Θέλουμε να έχουμε πάντα εμπειρογνώμονες και εκπαιδευμένους. Στα Ηνωμένα Έθνη ε, υπάρχει μεγάλη εμπειρία. Ξέρετε ότι θα ήταν σκόπιμο να υπάρχουν εμπειρογνώμονες σε θέματα ε, εργασιακά. Δεν υπάρχουν όμως πάντα. Τι ζητήσαμε στην Γενική Διεύθυνση ΕΜΠΛ αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η βιώσιμη ανάπτυξη, βιώσιμη. Αυτή είναι η λέξη κλειδί. Μιλάμε για βελτίωση του πλαισίου, αλλά νομίζω ότι το μέσον είναι πολύ καλό. Τώρα μπορούμε, πώς μπορούμε να το βελτιώσουμε. Έχει σημασία να ξέρουμε ότι είναι πολύ καλό το μέσον γιατί έγινε λόγος για το 2023 όταν λήξει το μέσον. Τι θα κάνουμε, θα το σταματήσουμε. Παρά την πρόκληση θα πρέπει να ξέρουμε τι θέλουμε. Εδώ έχουμε να κάνουμε με συγκεκριμένους τομείς που προσυπογράφουν οι ευεργετηθήσεις χώρες προωθούμε διεθνείς αξίες που δέχονται και οι ίδιοι δικαιούχοι μιλάμε για τα δικαιώματα των εργαζομένων, άρα οι χώρες θα πρέπει να τηρούν αυτά τα δικαιώματα. Ε, το GSP Plus πρόθυσε αυτούς τους διαλόγους. Υπήρχε η υποχρέωση, αλλά είναι καλύτερα να γίνεται διάλογος με κυβερνήσεις και μετά μπορεί να ανακύψει και κάτι άλλο. Όταν επισκέπτομαι αυτές τις χώρες, ξέρετε ότι προσπαθώ και προσπαθούμε να συναντηθούμε με εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών. Υπάρχουν χώρες όπου δεν υπάρχουν αρμονικές σχέσεις εμείς δίνουμε τις προτιμήσεις, δηλαδή το κίνητρο, το οικονομικό κίνητρο, αλλά αυτό θα πρέπει να οδηγήσει σε μια καλύτερη κατάσταση που θα αποτελέσει και feedback για μας. Πρόκειται για μακρύτερη διαδικασία. Άλλο είναι τα λόγια και ότι υπάρχει επιχάρτου και άλλο είναι οι πράξεις. Χαίρομαι για τις χώρες ε, δικαιούχος που είναι παρούσες γιατί μας δείχνουν ότι πραγματικά ε, έχουν δεσμευτεί. Γενικά νομίζω ότι αυτό που έχει σημασία είναι η δέσμευση θα πρέπει να υπάρχει δέσμευση και από εμάς αλλά και από τις χώρες. Θα ήθελα να ευχαριστήσω δημοσία το ΔΟΕ γιατί μαζί με το ILO μπορέσαμε να έχουμε ένα ανεξάρτητο σώμα εμπειρογνωμόνων πέρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ίσως να μην απάντησα σε όλες τις ερωτήσεις, αλλά όπως σας είπα δεν είχαμε οδηγίες χρήσης στην απαρχή του εγχειρήματο. Θα γίνει μια συνάντηση της κοινωνίας των πολιτών για την έκθεση Πρόκειται για μία πρόκληση που αφορά όλους τους συμμετέχοντες σε αυτή την αίθουσα. Σας ευχαριστώ πολύ όλους. Ελπίζω να παραμείνετε δεσμευμένοι. Ο κύριος Φιέλνερ έχει το λόγο. Ευχαριστώ και ευχαριστώ όλους τους ομιλητές που μας βοήθησαν να κατανοήσουμε καλύτερα το, πλαίσιο και την πραγματικότητα που διέπει αυτό το πλαίσιο και την έκθεση. Εμείς θα πάρουμε μαζί μας ιδέες για το πώς να συνεργαστούμε στα πλαίσια του GSP. Οι χώρες αυτές ε, δεν αφορούν πρότυπα τύπου Νορβηγίας, γιατί τότε δεν χρειάζονταν οι γενικευμένες προτιμήσεις. θα πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας στην πρόοδο. Ακούγοντας τη σημερινή συζήτηση θα πρέπει να διακρίνουμε ε, μεταξύ των 27 συμβάσεων και άλλων ανησυχιών και ζητημάτων που μας απασχολούν. Για παράδειγμα, η θανατική ποινή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ομόφωνα καταδικάζει τη θανατική ποινή. Αυτό είναι απόλυτα σαφές. Γι' αυτό μας ανησυχεί ιδιαίτερα όταν βλέπουμε ότι δεν τηρούνται. Θα πρέπει όμως να δούμε κατά πόσο θα πρέπει να υποστηρίξουμε προσπάθειες καταστολής της. θεωρήσαμε ότι οι γενικευμένες προτιμήσεις ε, δεν ε, αρκούν για να μας βοηθήσουν να καταπολεμήσουμε πάντα όλες τις ε, παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Θα πρέπει να δούμε τι γνώμη έχει, έχουν είπα ΙΠΑ, η Ιαπωνία και ούτω καθεξής. Έχουμε όμως και τομείς που καλύπτονται από τις 27 συμβάσεις και εδώ γνωρίζουμε ότι δεν μπορούν να επιληθούν όλα τα προβλήματα αλλά βρισκόμαστε στη σωστή οδό. Γι' αυτό και θα πρέπει να έχουμε μία πραγματική εταιρική σχέση όπου οι πάντες προσετερίζονται τις γενικευμένες προτιμήσεις. Υπάρχει κοινή προσέγγιση για την εφαρμογή των 27 συμβάσεων. Και εκεί έγκυται η αξία να τεθούν σε εφαρμογή οι γενικευμένες προτιμήσεις και αυτό το σύστημα. Πρέπει να είμαστε αυστηροί και να αποσύρουμε το GSP Plus εκεί που πρέπει. Δεν είναι κάτι το θεωρητικό. Έχει ε, συμβεί στο παρελθόν γιατί όταν αποσύρουμε αυτό το σύστημα τότε η εταιρική σχέση βοήθησε για να μπορέσουμε να επιτελέσουμε αυτή την πρόοδο μέσα στα πλαίσια των 27 συμβάσεων. Τέλος, πιστεύω ότι θα πρέπει να μας απασχολήσει το εξής. Μέσα στα πλαίσια των νομοθετικών αυτών πράξεων λέμε ότι σε τακτά χρονικά διαστήματα γίνονται αναθεωρήσεις. Στην περίπτωση αυτή το 2023. Πιστεύω λοιπόν ότι θα πρέπει να έχουμε κατά νου ότι το σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων συν θα πρέπει να έχει γερά θεμέλια για να δούμε πώς θα κινηθούμε μετά το 2023, έτσι ώστε όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς να έχουν απόλυτη εμπιστοσύνη σε αυτό το σύστημα και να μην υπάρχει ανασφάλεια. Ε, βεβαίως το 2023 φαίνεται μακριά, αλλά στην ουσία δεν είναι. Ich glaube, es ist ziemlich egal. Vielen Dank. Ευχαριστώ όλες και όλους που προσήλθατε σήμερα εδώ, που συζητήσατε μαζί μας. Και τώρα θα συνεχιστεί η συνήθις συνεδρίαση της Επιτροπής ΙΝΤΑ. Ο πρόεδρος Λάγκε, σας ευχαριστώ πολύ. Έμαθα πολλά από εσάς και τις παρεμβάσεις σας. Θα έρθουμε τώρα στο επόμενο θέμα της ε, Μηνεζίας Διατάξης, που είναι το υπαριθμό 18. Πρόκειται για την συζήτηση περί Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου και του θεματολογίου μετά τον Αερόμπι. Θα ήθελα να παρακαλέσω τον αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου Ας προσέλθει λοιπόν εδώ στο έδρανο του Προεδρείου καθώς και ο κύριος Αύσαν που είναι μέλος της Σουηδικής έρθει να καθίσει και αυτός εδώ δίπλα μας. Έχουμε πολλά μέλη της Steering Committee της Κοινοβουλευτικής Συνελεύσεως του ΠΟΕ εδώ κοντά μας και τους προσκαλούμε να συμμετάσχουν στη συζήτηση για την διαδικασία που αποκαλείται μετά τον αερόμπι. Όσοι επιθυμείτε να αποχωρήσετε Εάν θέλετε να συνομιλήσετε με τους διπλανούς σας, πράξτε το σιωπηλά. συνεχίζει ο πρόεδρος. Αγαπητές και αγαπητοί, έχουμε υπόψη το αποτέλεσμα της συνδιάσκεψης του ΠΟΕ στο Ναϊρόμπι. Είχα μάλιστα την τιμή να ηγηθώ αντιπροσωπείας 10 μελών του Ευρωκοινοβουλίου. Παρά τις περιορισμένες προσδοκίες που είχαμε στην αρχή και μέχρι το σχεδόν το τέλος η αισιοδοξία μας ήταν εξαιρετικά περιορισμένη. Εν τέλει βέβαια το αποτέλεσμα είναι ικανοποιητικό ακριβώς διότι υπήρξε αποτέλεσμα και η πολυμερής διαδικασία συνεχίζεται. Και όσοι είχαν προβλέψει το τέλος του ΠΟΕ τελικώς δεν δικαιώθηκαν. Άρα πρόοδος. Ούτε βέβαια μπορεί να πει κανείς ότι το αποτέλεσμα είναι τέτοιο που να δικαιολογεί κάποια ιδιαίτερη ισοδοξία. Είναι πάντως σημαντικό διότι προβλέπονται βήματα και σε αυτήν την ε, ατζέντα μετά τον Αϊρόμπι. Έχουμε μια ε, διακήρυξη που περιλαμβάνει διάφορα ενδεχόμενα βήματα που τελικώς ε, δεν αποδείχθηκε ότι μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο συνένεσης. Δύσκολο θα είναι βέβαια τώρα το καθήκον να προωθηθεί το περαιτέρω θεματολόγιο στη Γενέβη. Χαίρομαι που είναι παρόν ο αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής Μπράουνερ, έμπειρος άνθρωπος σε ό,τι αφορά την επιδίωξη συμβασμών, ήταν και εκπρόσωπος της Ομοσπονδιακής Γερμανίας στο TPC και έχει συμμετάσχει σε όλους τους γύρους διαπραγματεύσεων του ΠΟΕ από την Τόχα και μετά. Άρα όπως είπα είναι έμπειρος άνθρωπος. Θα σας δώσω τον λόγο και μπορείτε να μας εξηγήσετε πώς ε, νομίζετε ότι θα εξελιχθεί το θεματολόγιο μετά τον Αιρόβη. Σας ευχαριστώ. Επειδή με προσκαλέσατε ως εκπρόσωπο του ΠΟΕ και επειδή στον ΠΟΕ οι επίσημες γλώσσες είναι μόνο γαλλικά και αγγλικά θα μιλήσω αγγλικά. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου είναι ο οργανισμός ο οποίος διευθύνεται από τα μέλη του. Η γραμματεία λοιπόν δεν έχει δικαίωμα πρωτοβουλία. Δεν είμαστε όπω η Ευρωπαϊκή Ένωση όπου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαθέτει δικαίωμα ιδίας πρωτοβουλία. Δεν είμαστε εμεί εκείνοι που ορίζουμε την ημερήσια διάταξη του οργανισμού. Τα μέλη αποφασίζουν και τα μέλη βεβαίω επιφυλάζονται των δικαιωμάτων τους. Όπως γίνεται και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οποιαδήποτε λοιπόν πρόβλεψη σχετικά με το τι μπορεί να γίνει μετά τον αερόμπι δεν μπορεί παρά να λαμβάνει υπόψη το τι έχουν πει ή το τι ενδείξει έχουν δώσει ως τώρα οι χώρες μέλη. Δεν μπορεί να βασιστεί σε οποιαδήποτε δημιουργική προσπάθεια της γραμματείας. Την προηγούμενη Τετάρτη διεξήχθη η πρώτη ανεπίσημη συνάντηση των διαπραγματευτών μετά τον Αερόμπι. Πρόκειται για το όργανο το οποίο συνεδριάζει σε επίπεδο πρέσβεων. Ο επικεφαλής του οργάνου αυτού, ο Γενικός Διευθυντής, αντίλαξε απόψεις με τα μέλη. Ξεκαθάρισε ότι σύμφωνα με τη δική του εκτίμηση φύγαμε από τη Γενέβη για τον Αερόμπι με πολύ φτωχή προετοιμασία. Δεν είχαμε στους φακέλους μας ήδη συμπεφωνημένη υπουργική διακήρυξη. Όλες οι υπουργικές αποφάσεις και η ίδια η διακήρυξη βρίσκονταν σε μορφή σχεδίου και ακόμα πολλά πράγματα δεν είχαν συζητηθεί. Υπήρχαν πολλά ανεπίλητα θέματα τα οποία πήραμε μαζί μας για να τα πάμε στους υπουργούς αν μπορώ να το πω έτσι. Ο Γενικός Διευθυντής θεώρησε ότι ήταν αξιοθρύνητο αυτό και απέτησε από τους πρέσβει για τις μελλοντικές υπουργικές διασκέψεις να βελτιωθούν απαραίτητο οι προετοιμασίες. Τους απίφθινε έκκληση να βάλουν τα δυνατά τους, να σκόσουν τα μανίκια τους και να αναλάβουν περισσότερες πρωτοβουλίες. Δεν μπορούν να αφήνουν τις αποφάσεις να λαμβάνονται την 11η ώρα από τους υπουργούς επιτόπου. Οι πρωτεύουσε πρέπει να συμμετέχουν από νωρίτερα και μάλιστα και στι περιόδου μεταξύ δύο υπουργικών διασκέψεων. Ο Γενικό Διευθυντή τόνισε επίση ότι η διαδικασία του Ναϊρόμπι δεν ήταν ουδόλω ιδεώδη. Επέκρινε το γεγονό ότι πολύ συχνά δεν υπήρχε επαρκή διαφάνεια ούτε συμπερίληψη, inclusiveness. Έτσι, εν συνόψη, το πρώτο θέμα είναι για το μετά τον Ναϊρόμπι είναι αυτή η έκκληση του Γενικού Διευθυντού προς τους πρέσβεις να αναλάβουν περισσότερες πρωτοβουλίες και να είναι πλέον καλά προετοιμασμένοι για το μέλλον. Ο δίς από τα μέλη της ομάδας δεν αμφισβήτησε τις ε, κριτικές αυτές παρατηρήσεις του Γενικού Διευθυντού. Η Υπουργική Διάσκεψη στο Ναϊρόβι μπορεί να θεωρηθεί επιτυχία. Ωστόσο παρεβιάστηκε ένα ταμπού Ήδη το ανέφερε ο Πρόεδρός σας. Η Υπουργική Διακήρυξη στο τρίτο τμήμα της λέει καθαρά ότι υπάρχει μια ανεπίλητη ε, σύγκρουση μεταξύ των μελών. Με τον τρόπο αυτό η Υπουργική Διάσκεψη ξεφεύγει από την συνήθη προσέγγιση της αναζήτησης συνενέσεως και της συντάξεως ανακοινοθέντος στη βάση μιας ελάχιστης συμφωνίας. Στην διακήρυξη του Ναϊρόμπι αναφέρεται καθαρά η διαφωνία σχετικά με το μέλλον της DDA, δηλαδή της Doha Development Agenda. Ορισμένοι επιθυμούν να την εγκαταλείψουν λόγω του ότι δεν έχει επιτευχθεί καμία σημαντική πρόοδος τις τελευταία χρόνια. Γι' αυτό και με κάποια ανησυχία θα έλεγα εμείς από την πλευρά της γραμματείας αναμένουμε την πρώτη συνάντηση των Υπουργών στη Γενέβη μετά τον Αερόμπι δηλαδή, όπου θα φανεί καθαρά εάν αυτή η διαφωνία θα παραλύσει όλες τις μελλοντικέ διαβουλεύσεις. Η ανεπίσημη συνάντηση της Trade Negotiation Committee φαίνεται να δείχνει, να πάντως ότι αυτή η διαφωνία δεν θα κυριαρχήσει στις μελλοντικέ συζητήσεις. Όλα τα μέρη που έλαβαν το λόγο την προηγούμενη εβδομάδα ανεγνώρισαν ότι η έκβαση του Ναϊρόμπι είχε κάποια σημασία και του στο μέλλον θα πρέπει να συνεχιστεί. Από την, από, εξ αντιθέτου μάλιστα φαίνεται να είναι ξεκαθαρό ότι όλα τα μέλη συμφωνούν ότι τα ζητήματα της DDA, Doha Development Agenda, θα πρέπει να συνεχίσουν να συζητούνται ακόμα και αν τα μέλη της Επιτροπής διαφωνούν σχετικά με την αρχιτεκτονική των διαβουλεύσεων. Ορισμένα μέλη έθεσαν καθαρά την έμφαση στη διαπραγμάτευση νέων θεμάτων. Και αυτά τα μέλη όμως δεν αρνούνται να συζητήσουν θέματα της ίδιας της DDA. Σύμφωνα με την εκτίμηση του Γενικού Διευθυντού, όλα τα μέλη έδωσαν, ανέλαβαν μάλλον, να προωθήσουν, ανέλαβαν τη δέσμευση να προωθήσουν τις διαπραγματεύσεις για τα υπολοιπόμενα θέματα της ΔΟΧΑ. Είναι σημαντικό να το τονίσουμε αυτό, ακόμα και αν τα μέλη δεν συμφωνούν όλα για το πώς θα επιτευχθεί αυτό. Πρέπει να πει κανείς ακόμα ότι τα διάφορα μέλη έχουν δώσει διαφορετική έμφαση σε θέματα DDA ή για νέα θέματα. Ο Γενικός Διευθυντής ζήτησε από τους επικεφαλείς, από τους προέδρους να αρχίσουν συζητήσεις με τις οικίες διαπραγματευτικές ομάδες. Ένας αριθμός αντιπροσωπιών έθεσε νέα θέματα. Κανένα από αυτά όμως δεν έχει συγκεκριμενοποιηθεί το στάδιο αυτό. Γνωρίζετε βεβαίω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε με άλλες ευκαιρίες υποβάλει κάποια θέματα. Στην συνάντηση της περασμένης Τετάρτης δεν αναφέρθηκε ωστόσο κανένα συγκεκριμένο θέμα. Όπως είπα, ο ΠΟΕ διοικείται από τα ίδια τα μέλη του. Αναμένουμε λοιπόν τις ιδέες και τις ε, ε, αιτήσει των ίδιων των μελών εμείς της Γραμματείας. Η παρελθούσα εμπειρία δείχνει ότι τα μέλη εκείνα που επιθυμούν να συζητήσουν ορισμένα θέματα θα βρουν τρόπους για να το πράξουν. Είτε συμφωνούν όλοι, όλα τα μέλη δηλαδή με αυτούς, είτε όχι. Ελπίζω ότι οποιαδήποτε νέα διαβούλευση θα γίνει εντός του ΠΟΕ. Όμως υπάρχουν ενδείξεις ότι δραστηριοποιούνται έντονα κάποιοι και εκτός ΠΟΕ. Για παράδειγμα, Συμφωνία ΤΙΣΑ Ελπίζουμε ότι τα μέλη θα συμφωνήσουν επί των υπολοιπωμένων ζητημάτων DDA καθώς και θα βρουν τρόπο να συζητήσουν και τα νέα θέματα. Δύο υπουργικές διασκέψεις διαδοχικά επέφεραν κάποια πρόοδο. Έτσι λοιπόν οι επιχειρήσεις αρχίζουν, να ενδιαφέρονται και πάλι για το έργο του ΠΟΕ. Αυτό φάνηκε καθαρά και στο ε, Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός. Αναμένουμε λοιπόν από την επιχειρηματική κοινότητα να θέσει θέματα τα οποία να έχουν ε, σημασία. Ελπίζουμε ότι και εσείς ως εκλεγμένοι αντιπρόσωποι των λαών της Ευρώπης που ε, και από τις εκλογικές σας περιφέρειες γνωρίζετε πολύ καλά τα συμφέροντα και ενδιαφέροντα των εκλογέων σας θα μπορέσετε και εσείς να θέσετε παρόμοια θέματα. Θα ήθελα τώρα να κάνω και δύο πρόσθετες παρατηρήσεις για την Doha Development Agreement έχει δημιουργηθεί μια εξειδικευμένη διαπραγματευτική δομή. Υπάρχει δηλαδή η Trade Negotiation Committee, υπάρχουν και ξεχωριστές επιτροπές όπου συζητούν ζητήματα DDA. Κανένα από τα μέλη δεν αμφισβητεί την δομή αυτή. Ακόμα και τα μέλη εκείνα που επιθυμούν να εγκαταλείψουν την DDA δεν απαιτούν να διαλυθεί η δομή που ανέφερα. Αυτό είναι σημαντικό και δείχνει την καλή θέληση των μελών αυτών και επίσης συμβάλλει στο να αποφευθούν οι εσδήποτε περιπλοκές. Επιτρέπει δε και να υπάρξει μια πρόοδο στην διαδικασία. Έχω και μια άλλη παρατήρηση, ότι έχουμε μια ενσωματωμένη ατζέντα ή θεματολόγιο που προκύπτει από τις συμφωνίες ΠΟΕ που αναφέρονται στις συνεχιζόμενες διαπραγματεύσεις για γεωργία και υπηρεσίες. Εξάλλου, η διακήρυξη του Ναϊρόμπι ζητεί από τα μέλη, και αυτό συζητήθηκε στην προηγούμενη στη διάσκεψη, να συνεχίσει διαπραγματεύσεις για τον Special Safeguard Mechanism, να γίνουν διαπραγματεύσεις για επιτάχυνση του χρονοδιαγράμματος και να συνεχιστούν οι συζητήσεις για το βαμβάκι. Όλες αυτές οι δράσεις συνέχειας, follow-up, απαιτούν τώρα την προσοχή των μελών. Από την πλευρά της γραμματείας θα ήθελα να προσθέσω ότι υπάρχει ακόμη ένας αριθμός πολύ ενδιαφερουσών προσχωρήσεων που έρχονται, βρίσκονται στον αγωγό δηλαδή, και που έχουν τις δικές τους προκλήσεις. Βλέπε Λευκορωσία και Ιράν. Εν ώψη των πολλών διμερών ε, συμφωνιών ε, ελευθέρου εμπορίου που έχουν ε, ήδη γίνει αντικείμενο διαπραγματεύσεων καθώς και των ε, περιφερειακών συμφωνιών εμπορίου όπως η TPP. Η γραμματεία θα προβεί στην ανάλυση τους όταν θα έχουν, τις έχουν κοινοποιηθεί. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Είστε πραγματικός, αληθινός, γνήσιος διπλωμάτης. Είπατε κάποια πράγματα, βεβαίως αφήσατε και πολλά να εννοηθούν. Παρ' όλα αυτά η τοποθέτηση σας είχε ενδιαφέρον και θα ήθελα να προσκαλέσω τώρα τους άλλους συναδέλφους από την Διευθύνουσα Επιτροπή της Κοινοβουλευτικής Συνελεύσεως να λάβουν το λόγο. Πρώτος λοιπόν ο κύριος Αφσαν. Ευχαριστώ πολύ μόλις ξεκινήσαμε και να πω ότι από τη Διευθύνουσα Επιτροπή της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης για τον ΠΟΕ εκφράζουμε την ικανοποίησή μας. Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι που μπορούμε να πάρουμε μέρος σε αυτή τη συζήτηση. Ως Διευθύνουσα Επιτροπή είμαστε μια μεγάλη ομάδα των χωρών του ε, G20 συν και θα ήταν ε, μάλλον ε, όχι αρκετό να πούμε ότι πρέπει να συζητούνται οι περισσότερες πτυχές του εμπορίου ούτως ή άλλως. Ευχαριστούμε λοιπόν για τη δυνατότητα να πάρουμε μέρος και στην ακρόαση και σε αυτή την ενδιάμεση συζήτηση. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Άφσαν. Συνάδελφοι, μην διστάζετε, μην τρέπεστε να ζητήσετε το λόγο. Μπορεί να λάβετε κάποιες μη διπλωματικές απαντήσεις από τον ξέχοντα προσκεκλημένο μας. Πρώτη ερώτηση ο κύριος Μπίχνα. Ευχαριστώ που ήλθατε. Ερωτήσεις. Πώς αξιολογείτε την επίπτωση των πολιτικών δυσχεριών που φάνηκαν στον Αερόμπι για την επόμενη συνεδρίαση του Γενικού Συμβουλίου στις 24 Δευτέρου και πώς ποια πορεία θα ακολουθήσει ο ΠΟΕ μετά τον Αιρόμπι και πόσο ρεαλιστικό είναι να επιτευχθούν ακόμη σημαντικά βήματα πρόοδου. Και ένα εξειδικευμένο ερώτημα. Στη συμφωνία που επιτεύχθηκε στον Αιρόμπι για την Export Competition, ιδίω ό,τι αφορά τα γεωργικά προϊόντα, εκεί λέει στις παραγράφους 18 έως 21 ότι η δυνατότητα δυνατότητες κρατικών οργανισμών, αλλά ενδεχομένω και ιδιωτικών φορέων, είναι περιορισμένες. για να ορίσουν ελάχιστες τιμές ή να επηρεάσουν τις ελάχιστες τιμές για την εξαγωγή εμπορευμάτων. Ομιλεί και για μονοπωλιακές δράσεις. Βλέπω όμως μια ασυμμετρία η οποία οδηγεί τελικώς σε μειονέκτημα ή σε μειονεκτική θέση τους ίδιους τους αγρότες. Ο κύριος Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι αυτή η trade facilitation, διευκολύνση εμπορίου, είναι λοιπόν σημαντική πρόοδος και αυτή ήταν και η βάση για τον γύρο Τόχα και στο επίπεδο της Γεωργίας πετύχαμε ορισμένα πράγματα. Η ερώτησή μου τώρα αναφέρεται σε αυτό το Aid for Trade, βοήθεια έναντι εμπορίου. Είναι σωστό ότι η διάσταση αυτή μεταφέρθηκε στην COP21 και ότι τα Ενωμένα Έθνη θα το συνδυάσουν αυτό και με τον προβληματισμό για το διοξείδιο του άνθρακος και ότι θα μετακινηθεί αυτή η συζήτηση σιγά σιγά από τον ΠΟΕ στα Ενωμένα Έθνη. Θεωρείτε ότι το θεματολόγιο της ανάπτυξης θα επανέλθει στην επόμενη Υπουργική Συνάντηση, ο κ. Στάκουλα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ο πρώην διευθυντής του ΠΟΕ, ο κύριος Πασκάλ Λαμί, την περασμένη εβδομάδα δήλωσε σε μία διάσκεψη ότι οι διεθνείς οργανισμοί έχουν μία αποστροφή προς τις αλλαγές και ότι συχνά το πρόβλημα αυτό προκαλείται από την ηγεσία και το έλλειμμα στην ηγεσία. Μπορεί να υπάρχει κατακαιρματισμός, όμως κάποιος ηγείται στους διεθνείς οργανισμούς το γεγονό ότι δεν υπάρχει η κατάλληλη ηγεσία σε τέτοιο, σε τέτοιο διεθνής, διεθνές επίπεδο, κάποιο που να φέρει τι αλλαγέ και να τι υλοποιήσει, είναι ζωτική σημασία. Οι διεθνεί οργανισμοί είναι άκρως εξειδικευμένοι και κατακαιρματισμένοι στη λειτουργία του. Πρέπει κάποιο λοιπόν να συνδυάσει καλύτερα τι ε, δράσει του. Αυτό είπε ο κύριο Λαμί την περασμένη εβδομάδα. Επίση, είχε και τον ΠΟΕ κατά νου, πιστεύω, κάνοντα αυτό το σχόλιο. Ποιος λοιπόν είναι αυτός που πιλοτάρει τον ΠΟΕΣ σήμερα. Ο κύριος Αζεβέντο και οι διευθυντές του. Είναι ένας διεθνής οργανισμός που χρειάζεται ηγεσία. Το θέμα είναι λοιπόν ποιος θα αναλάβει να προωθήσει την πολυμερή ατζέντα. Και στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στον Ταβός η επίτροπο για την Οικονομική Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κυρία Μάλστρομ, είπε ότι πρέπει την πολυμερή ατζέντα να την διτηρήσουμε και να την προωθήσουμε. Υπάρχουν νέα ζητήματα, όπως το ηλεκτρονικό εμπόριο, το ψηφιακό εμπόριο, επενδύσεις και οι εγχώριες επιδοτήσεις. Αυτά λοιπόν μπορείτε να μας πείτε ποια μέλη του ΠΟΕ δεν θέλουν να συμπεριληφθούν ε, μεταξύ των προτεραιοτήτων Πώς θα μπορούσε να είναι μια πρωτοβουλία τη Ευρωπαϊκή Ένωση ρεαλιστική και να δοθεί συνέχεια. Υπάρχει κάποια άλλη πολυμερής πρόταση για αυτές τις ε, περιοχές δράσης. Ο κύριος Σόλτς. Ευχαριστώ πρόεδρε, ευχαριστώ για την απενημέρωση και για την δική σας αποτίμηση για το πώς έχουν πάει τα πράγματα τις πρώτες εβδομάδες μετά τον Αερόμπι. Είπατε ότι έσπασε ένα ταμπού. Από άποψη διαδικασίας τουλάχιστον. Πραγματικά μπορείτε να μου πείτε με κάθε ειλικρίνεια. Σημαίνει αυτή η ρήξη ότι υπάρχει κάποια συνένεση εντός του ΠΟΕ. Ότι στο μέλλον θα υπάρχει μια πιο διαθρωμένη προσέγγιση και εντός ΠΟΕ για τις διαπραγματεύσεις μεταξύ των διαφορών ομάδων χωρών. και στο πώς θα προασπίζονται τα δικά τους συμφέροντα. Θα προχωρήσουμε προς ένα σύστημα που είναι γνωστό και από άλλους παγκόσμιους οργανισμούς όπως ο ΙΕ για τις διαπραγματεύσεις και τους διάφορους γύρους διαπραγματεύσεων. Ποια θα ήταν η στρατηγική λοιπόν που θα ακολουθούσατε. Και δεύτερη ερώτηση. Το πρωί συζητήσαμε διαμακρόν τη θέση του Κοινοβουλίου για μια νέα διεθνή εμπορική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και δώσαμε έμφαση στις λεγόμενες global value chains, οι supply chains, τις ε, διεθνείς αλυσίδες παραγωγής. Αυτό θα εξαρτηθεί λοιπόν από τις δυνατότητες των εθνικών κρατών να διοργανώσουν τη δική τους οικονομική ανάπτυξη ανεξαρτήτως ή σε εξάρτηση με αυτές τις διεθνείς προεκτάσεις, διασυνδέσεις και διαπλοκές. Ε, είναι λοιπόν αυτές, ε, ποια είναι η άποψη του ΠΟΕ ως προς αυτό το στοιχείο. Είναι περιορισμένη η δυνατότητα δράσης σας. Και επίσης για τη συμφωνία Greenwood, ποια είναι η άποψή σας και πώς νομίζετε ότι θα μπορούσε να δοθεί συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ. Είμα. Ευχαριστώ Πρόεδρε, λυπάμαι γιατί δεν ήρθα εγκαίρως. Έπρεπε να παρευρεθώ σε άλλη συνεδρίαση που δεν είχε προβλεφθεί. Θα ήθελα να σας υποβάλω ορισμένες συγκεκριμένες ερωτήσεις. Καταρχήν, Ποια είναι τα βασικά διδάγματα ή συμπεράσματα, συμπεράσματα καθώς και οι βελτιώσεις του ΠΟΕ μετά την δέκατη υπουργική διάσκεψη, πώς μπορούν να βελτιωθούν τα δεδομένα και οι διαδικασίες. Επίσης, ποια είναι η άποψή σας για την παγκόσμια ε, εμβέλεια του ΠΟΕ. θα μπορούσε ο ΠΟΕ να ε, κατέχει πραγματικά η ηγετική θέση παγκοσμίω. Πώς μπορούμε να βελτιώσουμε την τεχνική αρρωγή στις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες έτσι ώστε να φτάσουμε σε συμφωνίες που πραγματικά να είναι ευεργετικές για τις χώρες αυτές. Τέλος, τι γνώμη έχετε για τις αναδιόμενες χώρες που κατά την άποψή μου έχουν αναδυθεί εδώ και πολύ καιρό και πώς μπορούμε να κατανείμουμε αυτές τις προσπάθειες για τις χώρες αυτές. Ευχαριστώ. Συνάδελφοι της ε, ε, Κοινοβουλευτικής Συνελεύσεως, έχετε και το δικαίωμα και το καθήκον να θέσετε ερωτήσεις. Ως τώρα δεν έχω κανέναν από τη δική σας πλευρά εγγεγραμμένο. Αλλά βεβαίως, όπως είπα, θα ακολουθεί ο κύριο και μετά εσείς που κάνετε νεύματα στο τέλος, στο βάθος εκεί. Ευχαριστώ κύριε αναπληρωτά γενική διευθυντά. Σας ευχαριστώ για την τοποθέτησή σας, βέβαια έχουν περάσει λίγοι μήνες. Νομίζω ότι ακόμη και αν οι γνώμες δίστανται και μεταξύ των Ευρωβουλευτών υπάρχει μια μεγάλη ε, πλειοψηφία υποστηρικτών του πολυμερού συστήματος. Υπάρχουν άλλοι που θέλουν ένα χαλαρό σύστημα. Ζητούμε να διατηρηθεί πάντως ζωντανό και δυνατόν και δραστήριο και φιλόδοξο στο στόχο του. Αυτή πάντως είναι η άποψη της πλειοψηφίας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο. Εδώ στην ε, Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου ε, έχουμε δεξαγάγει συζητήσει και πριν από τον Αιρόμπι, αλλά και ποιο μπορεί να είναι το μέλλον της ε, Doha Development Agenda και άλλα. Έχουμε συζητήσει και την διατλαντική σχέση. Αναμένουμε τώρα ότι ίσως να υπάρξει και TPP, θα δούμε. Πάντως ένα θέμα το οποίο επανέρχεται διαρκώς είναι το γεγονός ότι το δικαίωμα κύρωσης που διαθέτουμε μας αναθέτει και ευθύνες απέναντι στους ψηφοφόρους μας. Άρα χρειαζόμαστε ή επιβάλλεται διαφάνεια και ενημέρωση. Διαφάνεια και ενημέρωση σχετικά με, τις συγκεκριμένα, με τα συγκεκριμένα αποτελέσματα των προσπαθειών του ΠΟΕ. Και εκεί είναι το πραγματικό πρόβλημα, γιατί είναι πολύ δύσκολο να επικοινωνήσει κανείς για τα πράγματα αυτά με το κοινό και από την άλλη μεριά με... να αντιμετωπίσει κανείς τα επιχειρήματα αυτών που δεν πιστεύουν στο ελεύθερο εμπόριο. Δεν είναι εύκολο λοιπόν να προβάλλει κανείς επιχειρήματα υπέρ του εμπορίου. Όπως εξηγήσατε, όντως τα θέματα ε, του που τα, τα διαχειρίζονται τα μέλη του, δεν είσαστε όπως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο συνάδελφός μου πριν ανέφερε τον Πασκαλαμή. Είχε έρθει και πριν από ένα χρόνο νομίζω ο Πασκαλαμή, τον περασμένο Γενάρη ή Φλεβάρι εδώ, το 2015 είχε έρθει εδώ και είχε πει ότι μπαίνουμε στη νέα εποχή του εμπορίου, New Age of Trade, μπαίνουμε σε, σε καινούργιες ε, εποχές. Και αυτό περιλαμβάνει και αυτό το θέμα της επικοινωνίας. Είναι θέμα αυτό μέσα στα πλαίσια του ΠΟΕ. Θα ήθελα να ακούσω τις απόψεις σας. Ευχαριστώ πολύ. Ο συνάδελφός μας εκεί πίσω από την Κίνα. Ευχαριστώ Πρόεδρε, καταρχάς να ευχαριστήσω τον αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή του ΠΟΕ για την επινημέρωση. Ήταν και φωτιστική Ξέρουμε όλοι ότι η και τζάτα της Δόχας ε, κράτησε περίπου 15 χρόνια. Έχουμε πετύχει κάποια πράγματα, αλλά έχουμε και προκλήσεις και προβλήματα εντωμεταξύ. Σε αυτή τη φάση πρέπει να αντιμετωπίσουμε μια νέα κατάσταση που έχει διαμορφωθεί. Βρισκόμαστε σε ένα σταυροδρόμι, θα έλεγα, για το μέλλον. Όπως ανέφερε και ο αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή, κάποια από τα κράτη-μέλη θέτουν ένα βιβόλο και τις ίδιε του τι δεσμεύσει. Όπως ξέρουν όλοι, η Κίνα έχει την πεποίθηση, τη βαθιά πεποίθηση ότι το πολυμερές σύστημα εμπορίου είναι το καταλληλότερο. Γι' αυτό συμμετείχε ενεργά στην, ε, στους γύρους διαπραγματεύσεων της Δόχα. Σε αυτή όμως τη φάση δεν ξέρω. Είμαι μέλος του ε, εθνικού, ε, της Εθνικής Βουλής της Κίνας, του Λαϊκού Κοινοβουλίου της Κίνας, είμαι βουλευτής εκεί. Και θα ήθελα να μου πείτε στους συναδέλφους μου βουλευτές τι συμβουλή θα δίνατε ως αναπληρωτής διευθυντής του ΠΟΕ, πώς θα μπορούσαμε να στηρίξουμε την περαιτέρω ανάπτυξη και την συνέχιση της ανάπτυξης της πολυμερούς προσέγγισης, του πολυμερής, πολυμερούς εμπορικού συστήματος στο μέλλον. Ξέρουμε όλοι ότι οι διαπραγματεύσει αυτέ γίνονται μεταξύ κυβερνήσεων. Όμω, ω βουλευτέ, αυτό που μπορούμε να κάνουμε ίσω να έχει κάποια σημασία. Τι θα θέλατε εσεί να κάνουμε, λοιπόν. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε ο κύριος Ρούμπιχ. Δευτερολογία πολύ γρήγορα παρακαλώ. Η ερώτησή μου αναφέρεται στο market status που παρακολουθήσαμε και την προηγούμενη εβδομάδα. Εκεί για τη χαλιβουργία έχει μεγάλη σημασία, διότι για τους μικρούς προμηθευτές είναι ενδιαφέρον για να ε, μπορούν να λαμβάνουν σε χαμηλές τιμές ε, τα προϊόντα. Λάγε, υπάρχει κάποιος χρονικός ορίζοντας για να θεσπίσετε την ατζέντα σας και να την προωθήσετε. Και δεύτερο, υποστηρίζω την ε, κριτική του Γενικού Διευθυντού σας για την προετοιμασία των συνεδριάσεων διότι για την COP21 είχε δημιουργηθεί μια ομάδα ομοτήμων, ένα peer group που καθόρισε και το περιεχόμενο της ατζέντα. Δεν χρειάζονται άραγε κάποιες διαρθρωτικές αλλαγές στον τρόπο εργασίας και του ΠΟΕ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει και αυτή η ερώτηση για τον κ. Μπράουνερ. Όχι, έχετε το λόγο κύριε Μπράουνερ. Yeah, Σας ευχαριστώ πολύ, πολύ ενδιαφέρουσες οι ερωτήσεις και θα ήθελα να πω εξ αρχής ότι ε, εκτιμούμε το ενδιαφέρον του Κοινοβουλίου και βασιζόμαστε στην υποστήριξή σας. Αν δεν έχουμε την υποστήριξη τη δική σας και του επιχειρηματικού κόσμου, τότε δεν έχουμε παρά να αποχωρήσουμε. Παρακολουθούμε τι γίνεται, ποιες είναι οι εξελίξεις, οι εξελίξεις που προέρχονται από τα κράτη-μέλη. Άρα εσείς θα πρέπει να πιέσετε τις κυβερνήσεις και αυτό αφορά και τον Κινέζο επισκέπτη μας. Θα πρέπει να έχετε ε, την υποστήριξη του Κοινοβουλίου και το Κοινοβούλιο επηρεάζει την κυβέρνηση. Ο κύριος Μπούχνερ ρώτησε πώς θα προχωρήσουμε. Στο παρελθόν, όταν είχαμε πακέτα προς διαπραγμάτευση, το πρόβλημα ε, αφορούσε μια κατάσταση ομοιρίας. Είχατε ένα θέμα, υπήρχε ένα θέμα και ε, εάν ε, μάλλον οι, οι διαπραγματευτές προωθούσαν ένα ζήτημα, ανοίξαν ότι θα υπάρξει ένα αντίτιμο για παράδειγμα, όταν μιλήσαμε για το θέμα της ε, διαφάνειας στην ε, περίπτωση των διαδικασιών δύο αντιπροσωπείς είπαν δεν θα μιλήσουμε για τη διαφάνεια και τις διαδικασίες εκτός αν υπάρχει κάποιο αντάλλαγμα στον τομέα της γεωργίας. Αυτή είναι η κατάσταση ομοιρίας που ανακύπτει πολλές φορές. Άρα τώρα τα μέλη αποφασίσουν πώς μπορούν να αποφύγουν κάτι τέτοιο. Μπορούμε να το αποφύγουμε εάν διαπραγματευόμαστε ένα θέμα, κάθε θέμα ξεχωριστά. Ας πούμε η διευκόλυνση του εμπορίου ή τεχνολογίες πληροφοριών. Από μόνο του το θέμα, χωρίς συνοδευτικά σημεία. Ελπίζω τα μέλη να είναι αρκετά σοφά έτσι ώστε να μην ε, προβάλλουν προγράμματα όπου υπάρχει αυτή η ε, κατάσταση ομιλίας. Στη Βιέννη ε, με κάλεσαν οι αγρότες στην διεθνή τους διάσκεψη. Μιλούσαμε για την τον ανταγωνισμό στις εξαγωγές. Για την Ευρωπαϊκή Ένωση το θέμα αυτό δεν ε, ήταν ουσίας εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Η Ευρωπαϊκή Ένωση από το 2013 δεν έχει χρησιμοποιήσει καμία επιδότηση εξαγωγών και αυτό αφορά και τους αυστριακούς αγρότες οι οποίοι δεν ήταν δικαιούχοι τέτοιων επιδοτήσεων εξαγωγών παρότι πιστεύετε το αντίθετο. Ο κύριος Λαμή ε, εξέφρασε την απογοήτευσή του με βάση την ε, δική του εμπειρία. Ο ΠΟΕ κινείται από τα μέλη του. Και τώρα θα αναλάβω, θα πω κάτι το επικίνδυνο. Είχα πει και άλλες φορές ότι το 2013 από τον Οκτώβριο ε, βρίσκομαι σε αυτό το πλαίσιο εργασίας και προσπαθώ να δω ποιος είναι το ηγετικό ε, μέλος. Θα ήθελα να υπάρχουν περισσότερα κίνητρα στην οργάνωση. Υπάρχουν πολλοί οι οποίοι έχουν ε, ηγετική θέση, αλλά νομίζω ότι πολλές φορές χρειάζεται ουδέτερη στάση και να ζητήσουμε από τα μέλη να τα τι θέλουν να γίνει. Είναι δυσνόητο κάτι τέτοιο. Θα πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερο κίνητρο, μεγαλύτερη ε, όθηση, να δοθεί μεγαλύτερη όθηση στην οργάνωση. Και είπαμε στους πρέσβεις ότι θα πρέπει να ξεφύγουν από τα σημεία που τους διευκολύνουν. Θα πρέπει να έχουμε καλύτερη προετοιμασία. Και εάν δείτε στο Ναϊρόμπι, είχαμε πέντε χώρες που το τέλος ε, κατήχαν ηγετική θέση, αλλά μετά επικρίθηκαν διότι το θέμα της διαφάνειας δεν εντάχθηκε στη διαδικασία. Πάντα υπάρχουν συγκρουσιακές καταστάσεις, γιατί δεν μπορείτε να διαπραγματευτείτε παράλληλα με 164 χώρες και να έχουν όλη την ίδια πρόσβαση και διαφάνεια πάντα σε σχέση με αυτές που συμμετέχουν άμεσα σε ένα σχήμα και σε μία διαπραγμάτευση. Έχετε συμμάχους για τα νέα ζητήματα που ανακύπτουν. Βεβαίως ε, ισχύει κάτι τέτοιο, αλλά αυτή τη στιγμή δεν είναι σαφές πώς τα νέα αυτά ζητήματα που ανακύπτουν θα πρέπει να τύχουν διαπραγμάτευσης γιατί είναι πολύπλοκα ζητήματα και το ζήτημα είναι ποια πτυχή θα διαπραγματευτείτε στα πλαίσια του ΠΟΕ. Ο κύριος Σούλς υπέβαλε ένα ερώτημα. Βεβαίως η, συνένεση είναι το βασικό μας ενιολογικό πλαίσιο και οι διαπραγματεύσεις θα γίνονται εκεί που υπάρχει ενδιαφέρον και εάν δεν υπάρχει συμμετοχή ή αν δεν υπάρχει γενική συνένεση, τότε θα συνεργαστούν μικροομάδες. Οι Φιλιππίνες πάντα προωθούσαν τα θέματα των ΜΜΕ. Είναι ένα θέμα που δεν ήθελα να το συζητήσουν οι πάντες. Γι' αυτό θα δούμε πώς ε, ανακύπτουν τα πράγματα ως προς τα μέσα σε εξαγωγικά πράσινα αγαθά, green goods, θα ενταχθούν στο ολοπλαίσιο διαπραγμάτευσης και ελπίζω να επιτύχουμε και στη διαπραγμάτευση αυτή. Υπήρχαν πολλές ερωτήσεις ακόμα. σε σχέση με την ε, αλυσίδα αξιών. Αυτό το μελετήσαμε στο ΠΟΕ και στην ετήσια έκθεση του, του 13 νομίζω ασχοληθήκαμε με τα λεγόμενα value chains και εγώ επειδή ασχολούμαι με το πολύπλευρο εμπορικό σύστημα θεωρώ ότι τα value chains μπορούν να δημιουργήσουν ε, περίπλοκες απόρριες γιατί τα προϊόντα δημιουργούνται με βάση τα value chains και υπάρχουν και διμερείς ε, συμφωνίες μεταξύ των διαφόρων εταίρων και κάθε συμφωνία έχει τους δικούς της κανόνες. Όταν παράγεται ένα αγαθό μέσω αυτών των αλυσίδων Υπάρχουν πολλές διμερείς συμφωνίες που θα πρέπει να τηρηθούν καθ' όλη τη διάρκεια αυτών των ε, αλυσίδων και είναι πολύ δύσκολο να βρούμε από πού ανακύπτει αρχικά το ζήτημα. Και δεν έχει και ε, νόημα να δείξουμε και την προέλευση. Άρα κανείς αντιπαρέρχεται τις ε, προτιμήσεις για τις οποίες δημιουργήθηκε το αρχικό σχήμα. Άρα, με όλες αυτές τις διμερείς και περιφερειακές συμφωνίες και τους πολύπλοκους κανόνες προέλευσης, το ζήτημα θα επανέλθει στον ε, ΠΟΕ και θα υλοποιηθεί το, το, το πλαίσιο αυτό κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Άρα, τα value chains φτάνουν στα όρια που αναφέρατε, διότι το κάθε κράτος είναι κυρίαρχο μέσα στα πλαίσια της δικής του εταιρικής σχέσης, αλλά όχι καθ' όλη τη διάρκεια της, και εξέλιξη της αλυσίδας. Κύριε Βίνκλερ, υποβάλλατε ένα ερώτημα για το εμπόριο και τις ε, επικοινωνίες. Ναι, είναι ένα σοβαρό ζήτημα. Στην ε, κοινωνία των πληροφοριών είναι σαφές ότι το εμπόριο είναι ένα αξιόλογο μέσο για να απομακρύνει τους ανθρώπους από τη φτώχεια, και να τους κάνει πιο συμμετοχικούς σε μια, στην κοινωνία της επιμερίας, του πλούτου ας το πούμε έτσι. Όμως υπάρχουν πολλές επικρίσεις και κάθε χρόνο υπάρχει ένα δημόσιο φόρουμ που διοργανώνει ο ΠΟΕ και προσπαθούμε να δημιουργήσουμε μικρές ιστορίες εμπορίου για να δείξουμε πόσο πολλοί αντιπαρήλθαν ε, στη φτώχεια. Είχαμε πολλές μαρτυρίες από την Αφρική πέρσι. Θα έχουμε και άλλες τέτοιες εκπληκτικές ιστορίες από την Αφρική και τη Νοτιοανατολική Ασία για να δούμε ποια είναι η πραγματική συνεισφορά του εμπορίου. Σε σχέση με το καθεστώς της ε, οικονομίας της αγοράς είναι πολύ δύσκολο το θέμα Ως μέλος της γραμματείας δεν, ε, δεν έχω γνώμη. Αλλά ξέρω ότι το θέμα θα φτάσει στον ΠΟΕ. Όταν ένα κράτος μέλος προβάλλει μέτρα κατά της Κίνας και τότε η Κίνα θα παραπέμψει στο ζήτημα στο, σε επίπεδο δικαιοδοσίας και επίλυσης διαφορών του ΠΟΕ σε πρώτο επίπεδο και μετά θα φτάσει και στο ανώτατο επίπεδο. Θα απασχολήσει δηλαδή τον ε, ΠΟΕ μέσα στα πλαίσια ενός διακανονισμού, αλλά δεν μπορώ να λάβω θέση αυτή τη στιγμή. There Υπήρχε και το δικό σας ερώτημα για την τεχνική υποστήριξη και το ρόλο των αναδυόμενων χωρών οικονομίας της αγοράς. Ο ΠΟΕ βασίζεται στα μέλη του, άρα ε, κινούμαστε με βάση τη ζήτηση από τα κράτη και μετά προβάλλουμε προγράμματα τα οποία ανταποκρίνονται στο αίτημα του κράτους μέλους. Έτσι ώστε τα πλουσιότητα τέρα μέλη να παρέχουν τους σπόρους για να ανταποκριθούμε στο αίτημα αυτό, όπως ίσχυσε στο γύρο της Ντόχα. Ως προς αναδυόμενες χώρες αυτό είναι ένα από τα μεγάλα ζητήματα στον ΠΟΕ και τις ε, βιομηχανικές χώρες έχουμε τα LDC, τις ε, αναδυόμενες χώρες και ποιος θα πρέπει να είναι ο ρόλος αυτό των LDC, των λιγότερο αναπτυγμένων χωρών. Και αυτό ήταν ένα από τα βασικά θέματα της διάσκεψης του, του Ναϊρόμπι. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί το ζήτημα. Σας ευχαριστώ κύριε Μπράουνερ. Πολλές καυτές πατάτες όπως λένε στα αγγλικά μας δώσατε ή μάλλον έχετε εσείς στα χέρια σας. Σας εύχομαι καλή τύχη και κάθε επιτυχία στο έργο σας στην Γενέβη. Αγαπητές και αγαπητοί φίλοι, σας ευχαριστώ για την ενδιαφέρουσα συζήτηση και εσείς αγαπητοί φίλοι της ε, Διευθύνουσας Επιτροπής Steering Committee θα τα ξαναπούμε αύριο στις 10. Το επόμενο θέμα είναι η έκθεσή μας από τον Αερόμπι. Έχει διανεμηθεί, βρίσκεται και στην ιστοσελίδα μας, ο καθής μπορεί να το αναγνώσει. Το δε απολύτως τελευταίο είναι η ημερομηνία της προσεχούς συνεδριάσεως που θα διεξαχθεί στις 14 και 15 Μαρτίου. Σας ευχαριστώ πολύ και καλό σας βράδυ. Α, μη συγχωρείτε κύριε Τάκουλα, δεν σας είδα. Εξ όσων καταλαβαίνω, υπάρχουν και τα διάφορα. Α, τα αγαπημένο μου. Ναι, το ξέρω ότι το αγαπάτε ιδιαίτερα. Γι' αυτό αρπάζω την ευκαιρία. Πολύ γρήγορα. Επειδή χθε ήμουν στη Λαπωνία με την Επίτροπο Κρετσού δεν μπορούσα να παρευρεθώ στην συνεδρίαση και έγινε μια συζήτηση για τη Ρωσία. Είμαι μόνιμος εσύ για τη Ρωσία, όπως ξέρετε, σε αυτή την Επιτροπή και απογοητεύτηκα ιδιαίτερως όταν άκουσα ότι αναβλήθηκε η εξέταση του θέματος. Διότι στον Αρόμπι είδαμε το Ρώσο πρεσβή και νομίζω ότι είχαμε μια πολύ αποφελή συζήτηση. Νομίζω λοιπόν ο σωστός τρόπος να προάγουμε το, το ζήτημα θα ήταν να προσπαθήσουμε να γεφυρώσουμε λιγάκι τις διαφορές Ευρώπης, Ρωσίας και Ουκρανίας. Να μην δημιουργήσουμε νέα εμπόδια τώρα. Ελπίζω να επανέλθουμε λοιπόν στο ζήτημα αυτό και να βρούμε μια καταλληλότερη λύση. Να κάνουμε μια κίνηση προς τους Ρώσους, διότι αυτό που άκουσα χθε δεν ήταν, θα έλεγα, προσβλητικό, αλλά πολύ ευγενικό δεν θα το έλεγα. Ε, λοιπόν, απογοητευτικό το αποτέλεσμα. Αυτή πάντως είναι η δική μου προοπτική και η δική μου άποψη. Ο δικός μας ρόλος είναι να προσπαθούμε ως γιατροί να βρίσκουμε θεραπείες και να λύνουμε τα προβλήματα. Να βρίσκουμε λύσεις. Αυτό ήθελα να πω. να Ο, ο πρόεδρος Λάγκη, σας ευχαριστώ πολύ. Ίσως ορισμένα άλλα μέλη της ομάδας σας να μην έχουν την ίδια άποψη. Ε, ε, μπορεί να είναι και φήμη αυτό βέβαια. Ναι. Πάντως πράγματι επί της ουσίας έχει αναβληθεί το θέμα και θα το συζητήσουμε και θα πρέπει να βρούμε και το σωστό πλαίσιο για να το συζητήσουμε. Δεν έχω καμιά αμφιβολία γι' αυτό. Σας ευχαριστώ. Δεν έχουμε άλλα διάφορα. Καλό σας βράδυ.